Καλημέρα σας. Πριν αρχίσουμε τη συζήτηση, πρέπει να σας κάνω κάποιες ανακοινώσεις. Στα ρουμανικά θα το κάνω. Σε σχέση με τις αποφάσεις που έχουν λάβει διάφορες επιτροπές να αρχίσουν δύο οργανικές διαπραγματεύσεις, όπως ανακοινώθηκε την 3η 15η Ιανουαρίου, ο πρόεδρος δεν έλαβε έτοιμα ε, ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 69C παράγραφος 2 του κανονισμού. Συνεπώς, οι επιτροπές ΕΚΟΝ και Ήτρε... μπορούν να αρχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους. Αυτή ήταν η πρώτη ανακοίνωση. Και τώρα μπορούμε να περάσουμε στην ημερήσια διάταξη. Σύντομε παρουσιάσει των ακολούθων εκθέσεων. Πρώτα έχουμε την έκθεση του κυρίου Ντουγάν με θέμα τη διαφοροποιημένη ολοκλήρωση και του δίνω μέσω το λόγο για να μας κάνει μια παρουσίαση της έκθεσής του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την παρουσία σας. Έτσι νιώθω λιγότερο μόνος και μας και ε, την ψυχή ε, σήμερα το πρωί. Θέλω να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους ε, της Επιτροπής ΑΦΚΟ Συνταγματικών Υποθέσεων που είναι και παρόντες και ε, τον κύριο Χαουρεγγί και τους άλλους, ο οποίος κύριος Χαουρεγγί δεν εργάστηκε μόνο για την έκθεση αυτή αλλά και για τη δική του έκθεση γιατί η δική μου έκθεση για τη διαφοροποιημένη ολοκληρωσία εγγράφεται ε, στην ε, συνέχεια των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θυμάστε, είχε έρθει εδώ ο κύριος Γιούνκερ και παρουσίασε τα πέντε σενάρια. Ε, λοιπόν, είναι ε, στην τρίτη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία και προτιμά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μια Ευρώπη που προοδεύει και επιτρέπει και σε όσους θέλουν να προοδεύσουν και να πάνε παραπέρα να το πράξουν. Δεν χρειάζεται να επιμείνουμε σε αυτά τα θέματα. Ξέρετε ότι είναι ιδιαίτερε οι στιγμέ για την Ευρωπαϊκή Ένωση που ζούμε με το Brexit, με τη δυσκολία να ακουστεί η φωνή μας ε, από τους πολίτες και υπάρχει κίνδυνος να πέσουμε σε μια Ευρώπη πολλών ταχυτήτων. Πρώτη ταχύτητα για ορισμένους και για κάποιους άλλους δεύτερη, ακόμα και τρίτη ταχύτητα. Ε, όλη αυτή λοιπόν είναι μια πρόκληση που προσπαθούμε από κοινού να αντιμετωπίσουμε. Η έκθεση ε, ανοίγει κάποιες δυνατότητες και ενδεχόμενα και εντός συνθηκών και με προτάσεις για το μέλλον. Με κείμενες συνθήκες τώρα το Κοινοβούλιο επιμένει και θα επιμείνει πάρα πολύ για να χρησιμοποιούνται οι ρήτρες πασαρέλες λεγόμενες ε, για να φύγουμε από την εμπλοκή και την αγκύλωση. Θα πρέπει το πρωτογενές δίκαιο να ισχύει εξίσου για όλους. Και αν θέλουν να έρθουν και νέοι, ε, είτε θα υιοθετήσουν το σύνολο του πρωτογενού δικαίου, είτε θα περάσουμε από σε μια λογική εταιρική σχέση. Είναι πολύ σημαντικό οι συνθήκε να ισχύουν για όλε τι χώρε. Δεν υπάρχουν ε, διαφορετικά επίπεδα κρατών μελών ε, για το πρωτογενέ δίκαιο. Δεν νοείται κάτι τέτοιο. Πάρα πολύ σημαντικό για μα. Επίση, επιθυμούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να εδραιώσει ένα βάθρο θεμελιωδών δικαιωμάτων και να ισχύει και να μην υπάρχει η δυνατότητα η ε, υπαναχώρηση και οπισθοδρόμηση για τα θεμελιώδη δικαιώματα, ακόμα και αν είναι διαφοροποιημένη η ολοκλήρωση. Ε, για το τι μέλη γενέστε τώρα, θα θέλαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά να υπάρξει ένα πυλώνα κοινωνικών, περιβαλλοντικών, οικονομικών δικαιωμάτων ταυτόχρονα, έτσι ώστε να επιτρέψουν η Ευρωπαϊκή μα Ένωση να έχει μια ενιαία βάση και να προχωρεί με βάση αυτά τα θεμέλια. Αυτή είναι η γενική μα ε, προσανατολισμή. Κύριε Πρόεδρε, επιμένω θα πρέπει να φροντίσουμε η Ευρώπη να προχωρεί με μία φωνή σε ένα δρόμο, ε, όχι με πολλές ταχύτητες και ε, πολλές θέσεις και κατηγορίες, αλλά όσοι θέλουν να προχωρήσουν, να προχωρήσουν. Ευχαριστώ κύριε Λάινεν για το χειροκρότημα. Διαδικασία ΚΑΤΖΙΑΙ τώρα. Δύο συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Ο κύριος Μαριάς παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε καταρχάς να πω ότι το θέμα που συζητούμε είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον αλλά φυσικά δεν έχουμε την αναγκαία συμμετοχή. η ολοκλήρωση ούτως ή άλλως είναι διαφοροποιημένη σε επίπεδο ευρωπαϊκής ένωσης διότι έχουμε ε, τη σέγγεν στην οποία συμμετέχουν συγκεκριμένα κράτη μέλη ή την ευρωζώνη. Ω εκ τούτου λοιπόν είναι κάτι το οποίο γνωρίζουμε. δεύτερον έχουμε ορισμένα κράτη που έχουν πάρει εξαιρέσει με ειδικά πρωτόκολλα σε επίπεδο πρωτογενούς κοινοτικού δικαίου όπως είναι η δανία που εξαιρείται από συγκεκριμένες ρυθμίσεις ή επίσης η Ιρλανδία. Θα έλεγα λοιπόν ότι η ρύθμιση για τις χώρες που επιθυμούν να προχωρήσουν προβλέπεται πάλι μέσα ως διαφοροποιημένη ολοκλήρωση θεσμικά και επομένως είναι κάτι το οποίο πλέον εξαρτάται πολιτικά ποιες χώρες πρέπει να αξιοποιήσουν και αν θέλουν να αξιοποιήσουν αυτό το ζήτημα για να προχωρήσουν σε μια συνεργασία σε θέματα κοινωνικά ή περιβαλλοντικά θα έλεγα όμως ότι πρέπει να δούμε και το εξής ορισμένες χώρες λόγω ιδιαιτέρων προβλημάτων όπως είναι η ελλάδα η οποία ήταν μέσα σε μνημόνια όλα αυτά τα χρόνια δεν μπορεί εύκολα να συμμετάσχει επί ίσης με τους υπόλοιπους. γι' αυτό ίσως πρέπει να προβλέψουμε εντός της συνθήκης ορισμένες εξαιρέσεις για χώρες που έχουν μείνει πίσω ένα ειδικό καθεστώς I'm going to finish just a second, ένα ειδικό καθεστώς για ένα χρονικό διάστημα προκειμένου να μπορέσουν να ανακουφιστούν αυτές οι χώρες και να ακολουθήσουν τη διαδικασία ολοκλήρωσης στην πορεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η διαφοροποιημένη ολοκλήρωση είναι ένας ασαφής, συγκεχημένος και για το λόγο αυτό ε, δυσνόητος όρος με τον οποίο ορισμένα κράτη της ευρωπαϊκής ένωσης αλλά και κύκλοι της ευρωπαϊκής Ένωσης προσπαθούν να συγκαλύψουν ένα επικίνδυνο στόχο που έχουν θέσει για το μέλλον της ευρώπης δηλαδή την κατάργηση της σημερινής δομής της ευρώπης και την δημιουργία της ευρώπης των πολλών ταχυτήτων στην οποία θα έχει καταργηθεί η αρχή της ισότητας και ορισμένα κράτη θα είναι πιο ισχυρά από τα υπόλοιπα τα υπόλοιπα κράτη θα μετατραπούν σε παρείες θα τεθούν στο περιθώριο και εάν τους επιτραπεί θα συνεχίσουν την πορεία. η όλη κατάσταση μου θυμίζει τη γνωστή φράση από το έργο του Όργουελ, η φάρμα των ζώων ότι ορισμένα ζώα είναι, όλα τα ζώα είναι ίσα αλλά ορισμένα είναι πιο ίσα από τα άλλα. για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος πρέπει να καταργηθεί η αρχή της ομοφωνίας στη λήψη αποφάσεων της ευρωπαϊκής ενώσεως. με άλλα λόγια θα αποδυναμωθεί η ισχύ των κρατών και τα μικρά κυρίως κράτη δεν θα μπορούν να υποστηρίξουν τα συμφέροντά τους. επειδή αναφέρθηκα στον Όργουελ, θα κλείσω την παρέμβασή μου λέγοντας το εξής εάν δεν αντιδράσουμε σε αυτή την επικίνδυνη μεθόδευση τότε η ευρωπαϊκή ένωση είναι υποχρεωμένη να ζήσει το 1984 του Όργουελ και φυσικά να καταστραφεί. ευχαριστώ. Um, Κύριε Επιτίδη, δέχεστε γαλάζια κάρτα από τον κύριο Γιολάινεν. Παρακαλώ. Κύριε συνάδελφε, ε, ε, αυτό που λέτε τώρα είναι ότι όλα τα ζώα είναι τα ίδια ε, ορισμένα ίσα και κάποια άλλα είναι πιο ίσα. Υπάρχουν μεγάλα και μικρά κράτη. Θα συμφωνούσατε όμως όταν έχουμε 27-28 κράτη δεν μπορούμε πάντα να περιμένουμε μέχρι να ε, είναι όλα τα κράτη πρόθυμα ή σε θέση να κάνουν κάτι. Θα συμφωνήσετε ότι ορισμένα κράτη θα πρέπει να μπορούν να προχωρούν όπως έχει ήδη γίνει. Είναι μεν ανοιχτή η πόρτα για όλους. Αλλά όλα τα ζώα ε, είναι ίσα. Ορισμένα είναι πιο γρήγορα από τα άλλα και άλλα είναι πιο αργά. Αυτό είναι το θέμα. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Ε, όπως γνωρίζετε και όπως γνωρίζουμε όλοι η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζεται σε θεση να κανουν κατι θα συμφωνησετε οτι ορισμενα κρατη θα πρεπει να μπορουν να προχωρουν οπως εχει ηδη γινει ειναι με ενα ανοιχτη η πορτα για ολους αλλα ολα τα ζωα ειναι ισα ορισμενα αρχές και σε κάποιες αξίες ε, μία από τις αρχές αυτές είναι η αρχή της ισότητας η αρχή της ε, αλληλεγγύης η αρχή της συνεργασίας. άρα λοιπόν πρέπει σε αυτή την ένωση όλα τα κράτη να είναι ίσα και να συνεργάζονται μεταξύ τους. δεν πρέπει τα ισχυρότερα κράτη να επιβάλλουν την ε, θέλησή τους επί των υπολείπων. πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος συνεννοήσεως και συνεργασίας. υπάρχουν ορισμένα θέματα τα οποία αντιμετωπίζονται υπό το πρίσμα των συμφερόντων των μεγάλων κρατών και των ισχυρών κρατών. Αυτό δεν πρέπει να γίνεται. Τα μεγάλα κράτη δεν πρέπει να τεθούν στο περιθώριο. Ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Το λόγο τώρα έχει η κυρία Επίτροπος, η κυρία Γιωροβά. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, η έκθεση αυτή είναι μία ε, προσέγγιση που καλωσορίζουμε σε ό,τι αφορά και την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον και ε, προγραμματίζουμε λοιπόν ε, τις συζητήσεις μετά από το ΣΥΠΙΟ. Όπως ε, σημείωσε ο κ. Δουράντη, υπάρχουν διαφορές και όλοι ενδεχομένω κατανοούμε διαφορετικό τρόπο αυτή την διαφοροποιημένη ολοκλήρωση. Για κάποια κράτη-μέλη θεωρείται ότι είναι ένα θετικό βήμα προς την ενοποίηση αλλα κρατημέλη δε θεωρούν ότι προκαλείται κάποια σύγχυση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Λευκή Βίβλο σε ό,τι αφορά το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσίασε πέντε ενδεχόμενα σενάρια σε ό,τι αφορά τη συζήτηση. Το τρίτο σενάριο ήταν ε, να προχωρήσουν κάποιοι να δημιουργήσουν μια θετική ορμή προς την βαθύτερη ολοκλήρωση, ενώ άλλοι, όλοι μάλλον, να παραμείνουν ανοιχτοί για όσους έχουν διάθεση να προσχωρήσουν. Είδαμε με την πάροδο των ετών πώς ε, μπορεί να βοηθήσει αυτή η δυναμική για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις ε, και να προωθήσουμε την ε, ενοποίηση. Το ευρώ τώρα λοιπόν που γιορτάζεται 20 χρόνια του και η νομισματική ένωση καθώς και η ζώνη Σέγγεν αποτελούν παραδείγματα και μέσα σε τρία χρόνια είδαμε ότι όλα και πιο πολλά κράτη-μέλη εμπνεύστηκαν, θέλησαν να προσχωρήσουν σε τέτοιες ζώνες συνεργασίας. Ελπίζω και θεωρώ ότι το ίδιο θα συμβεί και για τη μόνιμη διατραμένη συνεργασία. Μια και τώρα οι Ευρωπαίοι πιο πολύ παραποτέ θα πρέπει να σταθούν ενωμένοι εν ώψη των... του πολιτικού σκηνικού στο παγκόσμιο προσκήνιο που αλλάζει. Υπάρχουν επίσης παραδείγματα και στον τομέα της δικαιοσύνης με την ε, δημιουργία για παραδείγμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το 2017 20 ήταν τα κράτη-μέλη τα οποία προσχώρησαν. 20 από τα 25 για τρια είχαν κάνει opt-out. 20 λοιπόν από τα 25 συμφώνησαν να ξεκινήσουν ενισχυμένη συνεργασία για να ιδρυθεί αυτή η βασική θέση για να καταπολεμηθεί η απάτη στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Έχουν προσχωρήσει έκτοτε και άλλα κράτη-μέλη και είμαι βέβαιη ότι σε τελική ανάλυση θα ακολουθήσουν και πιο πολύ. Αλλά η διαφοροποιημένη ολοκλήρωση αποτελεί μόνο μία δεύτερη, αν θέλετε, λύση. Η κανονική, η μέθοδος μέθοδο και η κανονική νομοθετική διαδικασία εξακολουθούν να αποτελούν τον καλύτερο τρόπο για να εγγυόμαστε την ακεραιότητα και την ευημερία του συνόλου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίση θα πρέπει να μείνει ανοιχτή η μορφή αυτή τη εργασία σε όλου όσου θέλουν να προσχωρήσουν. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρσι ξεκίνησε και συνεχίζει μάλιστα φέτο μια συζήτηση. Μια συζήτηση για μια πιο αποτελεσματική ε, διεξαγωγή διαλόγου και λήψη αποφάσεων για να γίνουν δυνατέ αυτέ οι αποφάσει, ε, όπω προβλέπεται και από τι ευρωπαϊκέ συνθήκε. Για την ε, ειδική πλειοψηφία σε κάποιου τομεί, όπω τι εξωτερικέ υποθέσει, τα φορολογικά, στο περιβάλλον. Αυτό θα επιλύσει και διάφορα μπλοκαρίσματα που προκαλούνται και θα οδηγήσει σε ενισχυμένη συνεργασία όπου η ομοφωνία δεν ε, είναι απαραίτητη και η ευρωπαϊκή δράση είναι κάτι που το επιθυμούν οι πολίτε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λοιπόν, προσβλέπει στην υποστήριξή σα ε, στα θέματα αυτά. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Επιτροπή, λέει ο Πρόεδρο. Και έτσι ολοκληρώνεται η συζήτηση και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα σήμερα. Και τώρα να περάσουμε στην δεύτερη έκθεση, στην ημερήσια διάταξη. Η έκθεση του κυρίου Λάινεν και της κυρίας Γιάννα Τούμ. Στρατηγική έρευνα τη διαμεσολαβητριά για τη διαφάνεια των νομοθετικών συζητήσεων στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το λόγο έχει ο, έχουν δύο εισηγητέ για τέσσερα λεπτά. Ο κύριο ε, Λάινεν, για να ξεκινήσει η συζήτηση, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε. Οι πολίτε ε, προσδοκούν οι αποφάσεις και κυρίως οι νομοθεσίες να είναι κατανοητές όλη η διαδικασία λήψη αποφάσεων να είναι διαφανή και κατανοητή. Αυτό το περιμένουν και οι πολίτε στα κρατημέλη, στι πατρίδε μα, αλλά το περιμένουν και από το επίπεδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί προφανώ απέχει πιο πολύ το επίπεδο το ευρωπαϊκό από τον πολίτη. Γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε ακόμα πιο πολύ διαφάνεια στο ευρωπαϊκό επίπεδο, πιο πολύ και από το εθνικό επίπεδο ενδεχομένω. Και το κοινοβούλιο αυτό αποτελεί ένα ανοιχτό κοινοβούλιο. Ό,τι ε, λαμβάνει χώρα στο κοινοβούλιο μπορούμε να το παρακολουθούν οι πολίτε. Ε, στο διαδίκτυο είναι ανοιχτέ οι συνεδριάσει μα, οι προπαρασκευαστικέ μα συνεδριάσει είναι ανοιχτέ. Είμαστε λοιπόν ένα από τα πιο διαφανή κοινοβούλια σε όλο τον κόσμο. Αυτό μα κάνει περήφανο. Αυτό δεν, συμβαίνει, δεν συμβαίνει όμως και στις άλλες, άλλες σώματα, στο Συμβούλιο Υπουργών, των 28 κρατών μελών. Εξακολουθεί να αποτελεί ένα μαύρο κυβότιο το Υπουργικό Συμβούλιο. Πολλά συμβαίνουν και κλεισμένα των θυρών. Έχουν βελτιωθεί βεβαίω τα πράγματα, αλλά απέχουν ακόμα παρασάγκα από το επιθυμητό επίπεδο. Πρέπει λοιπόν να απαιτήσουμε και το δεύτερο αυτό επίπεδο, το Υπουργικό Συμβούλιο, να διακατέχεται από πλήρη διαφάνεια όχι μόνο στην ψήφιση νομοσχεδίων, αλλά και στις 150 ε, προπαρασκευαστικές ομάδες που υπάρχουν, οι οποίες είναι απολύτως αδιαφανείς. Και ήταν πραγματικά κάτι το οποίο εκτιμήσαμε ιδιαίτερα από την διαμεσολαβητρία, το γεγονό ότι ε, ενέσκυψε το θέμα αυτό και εξέτασε όλα αυτά τα στοιχεία και τα αιτήματά μα. Εμεί λοιπόν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητούμε απόλυτη διαφάνεια στην, ε, στο δεύτερο σώμα λήψη αποφάσεων στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θα πρέπει πραγματικά οι συνεδριάσεις τους να είναι ανοιχτές, δημόσιες και προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις. Αυτό αντιτίθεται επίσης στην ε, τήρηση απόρριτων εγγράφων. Τα πιο πολλά ε, έγγραφα του Συμβουλίου έχουν τη σφραγίδα λεμιτέ, δηλαδή ε, απόρριτα. Ξέρουμε λοιπόν περιορισμένης ε, ε χρήσης. Αυτό δεν ήθιστε στις Βρυξέλλες. Είναι παροχημένο μέσο. Θα πρέπει λοιπόν το Υπουργικό Συμβούλιο να προσέχει πώς χρησιμοποιεί αυτό το μέτρο και να μην τα χαρακτηρίζει όλα να είναι πραγματικά πολύ λίγα αυτά τα έγγραφα, τα περιορισμένη ε, χρήση. Και συχνά οι υπουργοί έρχονται από τα εθνικά κράτη-μέλη αποφασίζουν ωραία ωραία κατά τι Βρυξέλλε και μετά λένε διαφορετικέ ιστορίε στι πατρίδε του. Και αυτό φυσικά μπορούν να το κάνουν, γιατί δεν υπάρχει κάποια απόδειξη του πώ έχουν ψηφίσει στο Υπουργικό Συμβουλίο. Και για εμά ω βουλευτέ και για του συναδέλφου στι εθνικέ βουλέ είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποφανθούν και να δηλώσουν πώ ψήφισε η εθνική κυβέρνηση. Μπορεί να βγαίνει ο καθένα να λέει ό,τι θέλει. Άμα θέλει το πιστεύει, άμα θέλει το πιστεύει. Ω εκ τούτου, λοιπόν, πιστεύω ότι η διαφάνεια στο Υπουργικό Συμβούλιο θα αποτελέσει και ένα μέσο καταπολέμηση όλων αυτών των θεωριών συνωμοσία. Έχουμε τόσου ε, λαϊκίστε ε, που φυσικά αρέσκονται στο να διαδίδουν τέτοιε ιστορίες. Νομίζω ότι έχει έρθει δεν πλήγαμε του χρόνου να δώσουμε αυτή τη διαφάνεια και να αποδείξουμε και να αποτελέσουμε και παράδειγμα, αν θέλετε, για τα κράτη-μέλη για την ε, καλή διαχείριση και την ε, καλή άσκηση διακυβέρνηση. Να ευχαριστήσω λοιπόν και τη συνάδελφα την κυρία Τούμ και όλου όσου ε, συνέβαλαν στην έκθεση αυτή και ελπίζω στι 12 η ώρα στην Ολομέλεια να ψηφίσουμε όλοι υπέρ τη έκθεση αυτή. Mm. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Λάινεν, λέει ο Πρόεδρο. Το λόγο έχει τώρα η κυρία ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, συνάδελφοι, Επίτροπε. Καταρχά, να ευχαριστήσω τη διαμεσολαβήτρια για τη δουλειά τη. Περίπου πριν από δύο χρόνια ξεκίνησε έρευνα για τη διαφάνεια στο Συμβούλιο και κατέληξε ότι οι τρέχουσε πρακτικέ στο Συμβούλιο δείχνουν ότι υπάρχει κακοδιαχείριση, ιδίω σε ό,τι αφορά την αδυναμία καταγραφή των θέσεων των κρατών μελών στι ομάδε εργασία, στι προπαρασκευαστικέ ομάδε του Συμβουλίου. Έκανε πολύ σωστέ συστάσει, όμω το Συμβούλιο δεν άκουσε. Απλώ δεν απάντησαν στην επιστολή τη, το φαντάζεστε. Γι' αυτό στράφηκε στο Κοινοβούλιο γιατί, για να έχει υποστήριξη. Στην πρώτη μα συνάντηση επί του θέματο, η Αυστριακή Προεδρία υποσχέθηκε να ασχοληθεί με το πρόβλημα ή τουλάχιστον να δώσει κάποια εξήγηση. Όμω η Αυστριακή Προεδρία απήλθε και δεν έχει υπάρξει ακόμα καμία απάντηση. Ελπίζουμε με τη Ρουμανική Προεδρία να αλλάξουν τα πράγματα. Η διαφάνεια στο Συμβούλιο έχει υπάρξει ένα θέμα συζήτηση εδώ και 25 χρόνια. Κι όμω δεν έχουν αλλάξει πολλά σε αυτό το διάστημα. Οι μικρέ νίκε που καταφέραμε, όπω την πρόσβαση στα έγγραφα των δημόσιων διαβουλεύσεων, που πίεσε για να τι έχουμε το Κοινοβούλιο και τη Διαμεσολαβήτρια, είναι ακόμα μικρέ. Πρέπει να έχουμε μεγαλύτερε αλλαγέ. Το Συμβούλιο ακόμα υποστηρίζει ότι η δουλειά του είναι πλήρω διπλωματική. Όμω η ε, φύση όλων των θεσμικών οργάνων έχουν αλλάξει με το καιρό. Ε, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο είναι συνομοθέτε. Θα πρέπει λοιπόν οι πρακτικέ που ακολουθούνται και στα δύο σώματα να είναι παρόμοιε. Το, το Κοινοβούλιο έχει γίνει πιο διαφανέ. Όλε οι συνεδριάσει επιτροπών, όπω ανέφερε ο Γιώργο Λάινεν, είναι ανοιχτέ και δημόσιε. Όλε οι θέσει είναι διαθέσιμε στο κοινό. Και οι θέσει του κάθε βουλευτή είναι ξεκάθαρε. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και το Συμβούλιο και τι ε, συνεδριάσει του Κορεπέρ πιο συγκεκριμένα. Θα πρέπει, όπω ε, λέγεται ξεκάθαρα στι συνθήκε, οι αποφάσει να λαμβάνονται όσο δυνατά πιο κοντά στο επίπεδο των πολιτών. Ιδίω τώρα, σε αυτέ τι ταραχώδει εποχέ του Brexit. Θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί ε, και όσο το δυνατόν κοντύτερα στους πολίτες. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα θεσμικά όργανα έχουν την υποχρέωση να είναι ανοιχτά στο κοινό και διαφανή. Είναι υποχρέωση όλων και είναι και καθήκον των συνομοθετών. Το κοινό περιμένει ένα αποτέλεσμα και ό,τι δεν πάει καλά, πολύ εύκολα τα κατημέλη το επιρρύπτουν στο κοινοβούλιο σε ευθύνη θα πρέπει να πάψει αυτή η διελκυστίνδα μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Ε, μερικά κράτη-μέλη έχουν πολύ ε, μετακίνητε θέσει και επιμένουν στι Βρυξέλλε σε επίπεδο Συμβουλίου. Αυτό είναι πρόβλημα για το Κοινοβούλιο, τα μέσα μαζική ενημέρωση και μετά τι Εθνικέ Βουλέ, που αργότερα ενημερώνονται για τι θέσει των κυβερνήσεών του, ε, αυτέ που έλαβαν στο Συμβούλιο. Εάν ενημερωθούν, πολλέ φορέ δεν ενημερώνονται καν. Αυτά τα σημεία τονίζονται στην έκθεση και ευχαριστώ τον Γιολάιναν για την καλή συνεργασία που είχαμε στην Επιτροπή. Και τέλο, να ζητήσω από το Σώμα να στηρίξει την έκθεση αυτή για να αποστείλουμε το μήνυμα ότι το Κοινοβούλιο θέλει διαφανεί δημοκρατικέ διαδικασίε. Ευχαριστούμε. Και τώρα η διαδικασία Κατσδιάη. Τέσσερι συνάδελφοι. Η κυρία Κινίτσι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η διαφάνεια της νομοθετικής διαδικασίας στην Ευρώπη είναι μια βασική συνιστόσα για να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Οι πολίτε θα πρέπει να μπορούν να ασκούν πλήρω το δικαίωμα ενημέρωσή του για τι εξελίξει τη ευρωπαϊκή νομοθεσία. Θα πρέπει να μπορούν να αναγνωρίσουν τις και να λάβουν γνώση των θέσεων των εκπροσώπων του. Είτε στο Κοινοβούλιο, είτε εμέσω με το τι συμβαίνει με τι κυβερνήσει και τι τοποθετήσει του στο Συμβούλιο. Οι Βρυξέλλε δεν μπορεί διαρκώ να απεικονίζεται από του κατηγορού τη ω ένα μαύρο κουτί, ε, το black box, όπου που μαγειρεύονται όπω θέλουν τα συμφέροντα. Θα πρέπει το καθήκον που έχουμε ω νομοθέτε για διαφάνεια να το ε, φέρουμε ει πέρα και να το σεβαστούμε. Η Επιτροπή ε, και το Κοινοβούλιο, όπω εντοπίζει η ίδια διαμεσολαβήτρια, έχουν κάνει σοβαρά βήματα για τη διαφάνεια στι προπαρασκευαστικέ του εργασίε τα τελευταία χρόνια. Είναι σημαντικό λοιπόν και το Συμβούλιο Συνομοθέτη να αναλάβει δεσμεύσει για να επιτύχει παρόμοια διοργάνωση στι πρακτικέ του, με τέτοια πρότυπα διαφάνεια βάσει των συστάσεων τη Ευρωπαϊκή Διαμεσολαβήτρια. Και επεξεργαζόμενο πρότυπα σαφή, ε, πολύ συγκεκριμένα για την ε, εμπιστευτικότητα των εγγράφων, όπω υπόθηκε μόλι τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο Μαριάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα το οποίο συζητούμε είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Το 1993 εξέδωσα ένα βιβλίο The European Ombudsman, στο οποίο είχα θέσει το ζήτημα της διαφάνειας και πώς ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής μπορεί να κάνει συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα θέατρο του παραλόγου. Το Συμβούλιο έχει δύο ρόλους. Είναι εκτελεστικό όργανο αλλά ταυτόχρονα είναι και όργανο νομοθετικό και όσο είναι όργανο νομοθετικό πρέπει να υπάρχει διαφάνεια πρέπει να γνωρίζουμε όλα τα προπαρασκευαστικά έγγραφα πρέπει να ξέρουμε κάθε κράτος μέλος τι λέει αναλυτικά πρέπει να γνωρίζουμε τι ψηφίζει κάθε κυβέρνηση. αυτό είναι σημαντικό για την άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου διότι ούτε οι βουλευτές στα εθνικά κοινοβούλια δεν μαθαίνουν τι ψηφίζει η κυβέρνησή τους. πολύ δε περισσότερο θα το γνωρίζουν οι πολίτες οι οποίοι στη συνέχεια θα κληθούν να ψηφίσουν τη συγκεκριμένη κυβέρνηση το συγκεκριμένο κόμμα ή να το καταψηφίσουν. άρα λοιπόν η έκθεση ανοίγει συγκεκριμένου δρόμου, η εργασία του ευρωπαίου διαμεσολαβητή είναι πολύ σημαντική για να υπάρχει επιτέλους διαφάνεια στο, συμβούλιο όπως υπάρχει διαφάνεια και στο κοινοβούλιο. να υπάρξει επίσης διαφάνεια και στο eurogroup διότι εκεί παίρνονται σημαντικές αποφάσεις που καθορίζουν την οικονομία και την πολιτική όλης της ευρωπαϊκής ένωσης. ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Η κυρία Άουκεν. Ευχαριστώ, ευχαριστώ τους δύο συγγητές. Ευχαριστώ και τη διαμεσολαβήτρια για την άριστη έκθεσή της. Εδώ βρισκόμαστε στο ε, στον πυρήνα της, ε, του δημοκρατικού ελλείμματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι το πρόβλημα ότι μιλάμε σε διαφορετικές γλώσσες. Το πρόβλημα είναι ότι οι εθνικές βουλές, τα εθνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν γνωρίζουν τι κάνουν οι κυβερνήσεις τους ε, και όλοι οι υπόλοιποι στις Βρυξέλλες. Φανταστείτε το κοινοβούλιο στη χώρα σας να, ε, να λέει ότι το κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες έκανε αυτό και εκείνο, υιοθέτησε το ένα και το άλλο, χωρίς να γνωρίζει καν τι συζητήσεις έγιναν στο κοινοβούλιο. Φαντάζομαι, περισσότερο δεν να πέσει αυτό. Όμως, ακριβώς έτσι εργάζεται το Συμβούλιο εργάζονται, λες και ήταν διακυβερνητικό θεσμό και όχι ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο με νομοθετικέ αρμοδιότητε. Με διπλωμάτε, με άλλε υπηρεσίε ε, και ευχαριστώ τη διαμεσολαβήτρια που το εντοπίζει αυτό στην έκθεσή τη. Ε, ελπίζω ότι θα πετύχουμε στήριξη για την έκθεση αυτή και θα πρέπει και στην προεκλογική σα εκστρατεία το θέμα αυτό να το προβάλλετε ω προτεραιότητα. Όλε οι κυβερνήσει πρέπει να ευαισθητοποιηθούν στο θέμα αυτό και έτσι μόνο θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι για το δημοκρατικό έλλειμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε. Ε, κυρία Άουκεν, δέχεστε καλά για κάρτα την κυρία Γκραπίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφε, Συμφωνώ απολύτως ότι δεν γνωρίζουμε αρκετά. Και μάλιστα αυτά που γνωρίζουμε δεν είναι και ακριβή πολλές φορές ε, για το Συμβούλιο. Οι πολίτες και τα κράτη, στα κράτη-μέλη δεν γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει. Ε, συχνά κατηγορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι τις κυβερνήσεις τους. Όμως πώς θεωρείτε ότι θα μπορούσαμε να τους πληροφορούμε καλύτερα τους πολίτες της χώρας μας για τις ευθύνες στο ευρωπαϊκό επίπεδο και για το τι πρέπει να γίνεται σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Εδώ υπάρχει αρκετή σύγχυση. Πολύ συχνά μάλιστα αυτό είναι θελημένο. Μιλάμε για η θελημένη σύγχυση που πολλέ φορέ προσκουρεί και στην αρχή τη επικούρικότητα. Δεν φταίνε μόνο τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ναι, εντάχει. Συμφωνώ, συμφωνώ. Αυτό προσπαθούσα και εγώ να πω. Ε, κυρία Γκραπίνη, πιστεύω ότι Εάν διαβάσει κανείς προσεκτικά την έκθεση της διαμεσολαβήτριας, αυτή που έχουμε μπροστά μα, ε, αναφέρει πολύ καλέ ιδέε για εργαλεία που επιτρέπουν να αντιμετωπιστεί σωστά το πρόβλημα. Τα εθνικά μέσα μαζική ενημέρωση, οι εθνικέ βουλέ, θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν καλύτερα τι κάνουν οι κυβερνήσει του. Θα αναγκάζονταν να δουν και την άλλη πλευρά του νομίσματο, δηλαδή τη νομοθετική διαδικασία, εδώ, στι Βρυξέλλε. Να παρακολουθούν τι κάνουμε εμεί. Δεν είναι λοιπόν το πρόβλημα μόνον ότι οι εθνικοί νόμοι εγκρίνονται εν αγνία. Είναι ότι σωστά πρέπει να ακολουθηθούν σωστά στις διαμεσολαβήτρια. Η κυρία Εύη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρώπη αυτή πολλέ φορέ δίνει την εικόνα ότι είναι απομακρυσμένη από του Ευρωπαίου πολίτε. Εάν μιλήσει κανεί με του απλού ανθρώπου, είναι σαφέ ότι η Ευρώπη ε, δεν είναι σαφέ ε, σε ποιον έχει αναθέσει να λαμβάνουν αποφάσει η Επιτροπή, το Συμβούλιο. Σωστά είπαν οι συνάδελφοι ότι το Κοινοβούλιο έχει μεγάλο βαθμό διαφάνεια στι εργασίε του. Όμω, όπω βλέπουμε, ε, πώ θα μπορούσαμε να πλησιάσουμε περισσότερο του Ευρωπαίου πολίτε, διότι ένα από τα τρία θεσμικά όργανα, το Συμβούλιο, ανέκαθεν εργαζόταν και, και κλεισμένο των θυρών. Και μάλιστα συμπεριφέρεται λε και ε, επιτρέπεται να παίζει ένα παιχνίδι πόκερ με κρυμμένα χαρτιά και πειραγμένη τράπουλα. Εδώ λοιπόν, ε, εδώ δεν είμαστε παίκτε, ούτε χαρτοπαίκτε. Στο Συμβούλιο έχουμε να κάνουμε με κράτη-μέλη. Γύρω από αυτό το τραπέζι ε, λαμβάνονται αποφάσει μείζωνο σημασία για το μέλλον των Ευρωπαίων πολιτών και τη ίδια τη Ευρώπη. Όλα αυτά λοιπόν καταπατούν τι αξίε τη ελευθερία και τη δημοκρατία και τι υποχρέωσει να ενημερώνονται οι πολίτε για τι αποφάσει που λαμβάνουν οι εκπρόσωποι του. Αυτό δεν μπορεί να αποδυναμώνει από το νόημά τη ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλουμε να απεικονίζεται με τέτοια άσχημη εικόνα η Ευρώπη στην ίδια την καρδιά τη. Ευχαριστούμε. Και τώρα η Επίτροπος Γιούροβα. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτέ, να σχολιάσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι αυτή η οποία θα σχολιάσει λεπτομερώ τι εσωτερικέ διαδικασίε που λαμβάνουν χώρα στο Συμβούλιο. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα ήταν δεσμευμένη να βελτιώσει τη διαφάνεια της νομοθετικής διαδικασίας εν γέννη, το οποίο αποτελεί κοινή ευθύνη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν ανέλαβε τα καθήκοντά της με τη δέσμευση να βελτιώσει τη διαφάνεια, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τους επιτρόπους, τα γραφεία τους και οι γενικές διευθύνσεις, οι γενικοί διευθυντές, ε, πάντα ε, συναντιόνται με τους ε, εκπροσώπους των επιχειρήσεων που είναι καταχωρισμένοι στο σχετικό μετρό διαφάνειας. Έχουμε λοιπόν αυτή τη διαφάνεια και ελπίζουμε και τα τρία θεσμικά όργανα θα συμφωνήσουν επί της συμφωνίας αυτής προκειμένου να υπάρξει μια γενική ένα γενικό μετρό για τους λομπιίστες. Επίσης, δημοσιεύουμε τις πληροφορίες για τις αποστολές αυτές, για τα έξοδα αποστολών, για τις συναντήσεις στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε επίσης υιοθετήσει νέους κανόνες για τους ε, συναντήσεις των εμπειρογνωμόνων, με ακόμα πιο αυστηρές προδιαγραφές για τα διαφάνεια. Και επίσης ε, δίνουμε χωρίς προηγούμενο πρόσβαση σε πληροφορίες σε ό,τι αφορά τις ε, διαπραγματεύσεις για ζώνες ελευθερού εμπορίου, τις διαπραγματεύσεις για το Brexit και βάσει λοιπόν της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο σας συμφώνησε για μια νέα διαθεσμική συμφωνία για την καλύτερη νομοθεσία, το οποίο θα περιλαμβάνει και μια κοινή δέσμευση βελτίωσης ε, της διαφάνειας της νομοθετικής διαδικασίας συμπεριλαμβανομένης και τη διάσταση των τριμερών διαπραγματεύσεων και την επικοινωνία με το ευρύ κοινό. Όπω σημειώνεται και στην έκθεσή σα, συνεχίζονται οι εργασίε μεταξύ των υπηρεσιών των τριών θεσμικών οργάνων για την ανάπτυξη κοινού νομοθετικού κόμβου που δεσμευτήκαμε να ιδρύσουμε. Θα είναι ένας τρόπος φιλικό προ το χρήστη για άτομα που δεν είναι ειδικοί να έχουν πρόσβαση παρόλα αυτά σε πληροφορίε σε ό,τι αφορά την τρέχουσα νομοθετική διαδικασία και πολλέ πληροφορίε διατίθενται ήδη. Αν γνωρίζει κανεί, φυσικά πρέπει να κοιτάξει. Αλλά αυτό φυσικά δεν είναι εύκολο πάντα. Δεν είναι εύκολο για του ανθρώπου ανθρώπους που δεν είναι ειδικοί. Αλλά μέσω του κόμβου αυτού θέλουμε να αλλάξουμε ακριβώ αυτό το στοιχείο. Αν λοιπόν το Κοινοβούλιο επιθυμεί να δημοσιεύει επιπρόσθετες πληροφορίες σε σχέση με αυτά που δημοσιεύονται, εκεί θα μπορούσε να το πράξει αυτό, σε αυτόν τον κομβό, τον δικτυακό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την Επιτροπό, λέει ο Πρόεδρος. Και έτσι ολοκληρώνεται η συζήτηση και θα λάβει χώρα ψηφοφορία σήμερα σε ό,τι αφορά την ε, άλλη έκθεση. Να καλώς ορίσουμε την Επιτροπό. Μάλμστρομ, η οποία μόλις ήλθε για το επόμενο θέμα στην ημερησία διάταξη, που αφορά τις περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Η πρώτη λοιπόν έκθεση για το Αζερμπαϊτζάν και συγκεκριμένα η υπόθεση του Μέχμαν Χουσέινοφ. και να δώσω το λόγο στη Ρεμπέκα Χάρμς για να σας καλωσορίσω κιόλα Να πάρετε το λόγο, παρακαλώ. Ε, ε, Ευχαριστώ. Καλημέρα σας, κύριε Επίτροπε, κύριε και κύριοι. Χαιρετώ και όσους στο Αζερβαϊτζάν ενδεχομένως να παρακολουθούν τη συζήτηση. Αζέρι Daily είναι μια διαδικτυακή εφημερίδα όπου διάβασα ένα άρθρο ε, και εγώ και οι συνάδελφοι ε, που δουλέψαμε για το ψήφισμα αυτό κατηγορούμαστε ότι συνομωτούμε στην προετοιμασία πραξικοπήματος κατά της κυβέρνησης της χώρας. Συνιστώ στους δημοσιογράφους αυτής της εφημερίδας να μας ρωτάνε, να συζητάνε πριν γράφουν τέτοια πράγματα θέλω να απευθυνθώ και στους συναδέλφους μου, ε, τους βουλευτές του Αζερβαϊτζάν που τους γνωρίζω ε, ε, από την Euronest. Δυστυχώς δεν κατάφερα να τους δω να συνεννοηθώ μαζί του. Ο Φουάτ Μοράντοφ, τον οποίο γνωρίζω από παλιά και ήταν συνάδελφος, είναι πλέον υπουργό στην κυβέρνηση του Αλίεφ και ξέρει ότι ανέκαθεν στη συνέλευση Euronest ε, εγώ ε, ήθελα να έχουμε καλές σχέσεις και σχέσεις εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας οι βουλευτές. Γιατί παρουσιάσαμε αυτό το κατεπήγον ψήφισμα και το γράψαμε στην μερίσια διάταξη. Ανησυχούμε για τη μοίρα του Μεχμέαν ε, Χουσεϊνοφ ο οποίος κρατείται από πέρσι το Δεκέμβριο και μάλιστα κάνει απεργία πείνας από τον περσινό Δεκέμβρη διότι τον απειλούν πριν λήξει η ποινή του που έχει καταδικαστεί σε δύο χρόνια φυλάκιση ε, του απαγγέλθηκαν και νέες κατηγορίες και τώρα φοβάται ότι θα του επιβληθεί και άλλη ποινή 5 με 7 έτη ε, φυλάκισης πριν λήξει καν η προηγούμενη ποινή του. Η κατάσταση αυτή δεν είναι καθόλου μεμονωμένη. Το Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών ε, στην κοινοβουλευτική συνέλευση Euronest μας ε, ενημέρωσε ότι αυτή η κατάσταση επαναλαμβάνεται ως ε, σχήμα για πέμπτη φορά. Και Ακριβώς γι' αυτό το λόγο καταθέσαμε και γράψαμε στην ημέρη σε διάταξη το συγκεκριμένο ψήφισμα. Όλες οι πολιτικές ομάδες απευθύνουμε έκκληση στην κυβέρνηση του Αζερβαϊτζάν να αφήσουν ελεύθερο τον Μεχμάν Χουσέινοφ. Απευθύνουμε έκκληση και στους δικαστές να μην επιτρέπουν τέτοια σκηνοθετημένα ε, σχήματα. Ο Χουσέινοφ αποκάλυψε τη διαφθορά στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Γι' αυτό τον έχουν φυλακίσει. Και δεν έχει ασχοληθεί μόνο με τα προβλήματα που υπάρχουν στο Αζερβαϊτζάν, αλλά και άλλα προβλήματα με διεφθαρμένους πολιτικούς, παράδειγμα στη Γερμανία και στην Ιταλία. Και γι' αυτό το λόγο είναι σωστό που ασχολείται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ζητεί την άμεση και άνευ όρων αποφυλάκησή του. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ο κύριος Κοράου. Δύο λεπτά. Thank you, Mr. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα σας, Επιτροπή. Φαίνεται ότι δεν υπάρχουν πλέον ε, σύνορα για τον Πρόεδρο Άριεφ. Το μήνυμα αυτού του δικτατορία είναι σαφές. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να εκθέτει την ε, διαφθορά και τι εκτεταμένε παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αξιωματούχων του Αζερβαϊτζάν και τη κυβέρνηση. Ο κ. Χουσέινοφ είναι εμβληματική περίπτωση. Ο blogger αυτό έχει ε, παρενοχληθεί από την αστυνομία επί σειρά ετών και μετά ε, φυλακίστηκε αφού συνελήφθη και βρίσκεται στην ε, βρίσκεται στη φυλακή. Εδώ προσπαθούν να φημώσουν μια από τις φωνές που προασπίζεται τα ανθρωπινά δικαιώματα στο Αζερβαϊτζάν έχει τύχει κακομεταχείριση βασανιστήριων και κατηγορήθηκε για δυσφήμιση των ίδιων των αξιωματούχων που τον βασάνισαν. Ε, τι θα μπορούσε να κάνει όμως μια χώρα όπου είναι 136 της 180 χώρες στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τι περιμένετε για τους δημοσιογράφους και ε, τους blogger ε, που δεν θέλουν να υποκύψουν ε, στους εκβιασμούς, τις, τα βασανιστήρια και τους ξυλοδαρμούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται για νέα συμφωνία με το Αζερβαϊτζάν. Θα έπρεπε να βασίζεται στο διεθνέ δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την καλή διακυβέρνηση και τι δημοκρατικέ μεταρρυθμίσεις. Οι αρχέ αυτέ όμω δεν πρέπει να παραμείνουν μόνο λόγια στο χαρτί. Θα πρέπει μελλοντικέ συμφωνίε του Κοινοβουλίου ε, να μην ε, συνάπτονται, παρά μόνο αν αλλάζει δραστικά η κατάσταση στη χώρα κατάσταση αυτή στο Αζερβαϊτζάν, η κατάσταση αυτή υποβάθμιση των δημοκρατικών δικαιωμάτων πρέπει να αλλάξει. Και θα πρέπει η απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων να γίνει προτεραιότητα και στη δική μα πολιτική. Θα πρέπει να ασκήσουμε πίεση στι αρχέ του Αζερβαϊτζάν για να αποσύρουν τι κατηγορίε και χωρί όρου να αποφυλακίσουν και τον κύριο Χουσέινοφ και του άλλου δημοσιογράφου που βρίσκονται στη φυλακή. Εάν δεν γίνει αυτό, θα προσπιστούμε τι αρχέ και τι αξίε μα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριο Στάνοκ για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ε, εδώ και δύο χρόνια περίπου ο Μεχμάν Χουσέινοφ καταδικάστηκε σε διετή κάθριξη για ε, υποτιθέμενη δυσφήμιση. Προσπάθησε απλώς να εκθέσει τη διαφθορά των κυβερνώντων στη χώρα του. Και ανέκαθεν ε, υπήρχαν υποψίες ότι όλες οι κατηγορίες αντίον του ήταν πολιτικού χαρακτήρα. Με τη δίκη του να πλησιάζει, οι αρχές προσπαθούν τώρα να εξαγγείλουν νέες κατηγορίες ώστε να πετύχουν ποινή εξαετή ή οχταετή. Και φυσικά είναι αβάσιμες οι κατηγορίες αυτές. Ε, ήδη υπάρχουν φήμες ότι αυτό το μήνα μόνο προκύψαν πέντε τέτοιες επιθέσεις παρόμοιες με ψευδείς κατηγορίες για φυλακισμένους των οποίων οι ποινές πρόκειται να ε, λήξουν κάπου τώρα. Θα πρέπει λοιπόν ε, να δούμε και τη θέση του Αζερβαϊτζάν, που είναι 163η χώρα από τι 180 χώρε για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι από τι χειρότερε επιδόσει στον κόσμο. Θα πρέπει λοιπόν η υπόθεση αυτή να συζητηθεί σήμερα εδώ, να τονιστεί και δεδομένη τη ε, κακή υγεία του κ. Χουσέινοφ, που είναι, κάνει απεργία πείνα, ε, να γίνει κάτι, να πιέσουμε για την άμεση απελευθέρωσή του και αρχές να πάψουν την εξαγγελία κατηγοριών ε, στο Αζερμπαϊτζάν, μια χώρα της Ανατολικής Γειτονίας που συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με την οποία έχουμε καλέ σχέσει. Ε, Ο κ. Ουρμπάν Κρέσπο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στο Αζερβαϊτζάν η διαφθορά δεν είναι ένα κάποιο πρόβλημα είναι ενδυμική και όποιος τολμάει να την καταγγείλει ε, καταλήγει στη φυλακή όπου το βασανίζουν και όλος. Αυτό συζητούμε τώρα αυτή τη στιγμή. Ε, και είναι η κατάσταση του Μεχμάν Χουσεϊνοφ που έχει καταδικαστεί σε διετή φυλάκιση και τώρα κινδυνεύει και με άλλα 7 έτη. Το 2017 πριν ε, τον συλλάβουν είχε ξεκινήσει μια εξτρατεία κατά της διαφθοράς της ελίτ που κυβερνάει στο ε, Αζερβαϊτζάν. Είχαν βρει μια μυστική ε, κομπίνα για να πληρώνουν Ευρωπαίους να αγοράζουν πολυτελή ε, κατοικίες και να ξεπλένουν χρήμα. Όλα αυτά εξαγόρασαν Ευρωπαίους πολιτικούς και δημοσιογράφους για να μην επικρίνουν τον πρόεδρο, για να φημώνουν ε, όσους καταγγέλουν ε, τη βαραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για να προωθούν την, ε, μια ωραία εικόνα για τη χώρα. Αυτό ονομάστηκε η διπλωματία του Χαβιαριού. Ο Πέντρο Αγγραμούν ήταν ένας από εκείνου που χρειάστηκε ε, να παρετηθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης, από τα ε, αξιώματά του μετά από αυτά τα σκάνδαλα. Αλλά επειδή φαίνεται να ενδυμεί και στο κόμμα του το ίδιο, ε, το Λαϊκό Κόμμα παραμένει γερουσιαστής στην Ισπανία. Υπάρχουν μεγάλα έργα στο Αζερβαϊτζάν, είναι πηγή φυσικών πόρων, ε, ενεργειακός προμηθευτής για να ξεφύγουμε από την εξάρτηση ε, στην Ρωσία. Από εκεί ξεκινάει ε, πέτρελαιο και αγωγός φυσικού αερίου. Πάνω από 1.700 χιλιόμετρα μεταφέρει ο αγωγός πετρέλαιο στη Δύση. Η BP, British Petroleum, πριν από 10 χρόνια ε, άρχισε αυτή την προσπάθεια για να ξεπλύνει την εικόνα του Αζερβαϊτζάν στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Θέλουμε να ε, ματαιωθεί ε, οποιαδήποτε ευρωπαϊκή συμμετοχή στο διάδρομο του Νοτιού Καυκάσου, να σταματήσουν οι διαπραγματεύσεις γιατί δεν θέλουν να σέβονται καθόλου την ελευθερία της έκφρασης του συνέρχεστε και του συνεταιρίζεστε στη χώρα τους. Πριν από λίγους μήνες αποφασίσαμε να βάλουμε όρους στη συνεργασία μας για την κοινωνία των πολιτών και τους φυλακισμένους πολίτες. Ακόμα περιμένουμε. Το 2017 ζητήσαμε να διερευνηθεί το θέμα αυτό, η απάτη, η καταπολέμηση ε, της διπλωματίας του Χαβιαριού δεν έχει προχωρήσει. Και ζητούμε από τις Ισπανικές αρχές να χρησιμοποιήσουν όλους τους μηχανισμούς που έχουν για να διερευνήσουν ε, αυτές οι κατηγορίες κατά του γερουσιαστού Πέδρο αδραμούν και να τον ε, κάνουν να παραιτηθεί. Για άλλη μια φορά πρόκειται για εξωτερική πολιτική της Ένωσης με τους γείτονές της. Πού είναι οι αρχές και οι αξίες. Διαπλέκονται με τα συμφέροντα και δεν μπορούμε να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις αν δεν ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας και αν δεν βάλουμε όρους και προϋποθέσεις στη συνεργασία με το Αζερβαϊτζάν. Κύριε Σχάκε, για τρία λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και καλημέρα στην Επίτροπο. Καλημέρα στην αδελφή. Είναι λυπηρό το γεγονό ότι βρισκόμαστε και πάλι εδώ και συζητάμε την επιδείνωση των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αζερβαϊτζάν. Υπό την ηγεσία του ε, Πρόεδρου Αλιεύ και τη αντιπρόεδρου, τη γυναίκα του. Και ο, η περιπτώση του κ. Χουσονέφα ε, δείχνει τι γίνεται σε ό,τι αφορά την παράνομη κράτηση του, τα βασανιστήρια που υπόκειται και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία, το κράτο δικαίου παραβιάζονται συστηματικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμω ε, αυτό το καλοκαίρι υπέγραψε συμφωνία ε, συνεργασία με το Αζερβαϊτζάν. Θα πρέπει να κοιτάξουμε την αρισιμότητα και πώ μπορούμε να την αξιοποιήσουμε. Γιατί κάθε συμφωνία σύνδεση με οποιαδήποτε χώρα δεν μπορεί να αποτελεί λόγο ή δικαιολογία για να αποφεύγουμε την ε, επισήμανση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τους πιο αυστηρούς όρους. Και το Αζερβαϊτζάν είναι στη θέση 163 από τις 180 χώρες σε ό,τι αφορά την ε, παγκόσμιο δίκτυ για την ελευθερία. Είναι πραγματικά σοκαριστικό το γεγονός αυτό και μιλάμε για άτομα τα οποία είναι σε φυλακή, μιλάμε για ε, κάποια website και blog στις χώρες και τα πιο λαμπρά μυαλά της χώρας έχουν ήδη διαφύγει γιατί ουσιαστικά διακυβεύεται η ζωή τους και των οικογενειών τους. Όπως είδαμε λοιπόν διαρροές, δειλές ε, τέτοιων βίντεο και 23.000 ευρώ της κυρίας Ισμαήλοβα. Μιλάμε το δεκαπλάσιο του ετησίου εισοδήματος της χώρας. Αυτό καταδεικνύει πόσο πίεση ασκείται στους δημοσιογράφους, αλλά και η πίεση που ασκείται στους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης. Η συνολική κατάσταση σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιωμάτα είναι πολύ δεινή. Φυλακίσεις, εκφοβισμοί και φυσικά έμεση παραβίαση των υποχρεώσεων του Αζερβαϊτζάν από την υπογραφή της συνθήκης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όταν λοιπόν θα κοιτάξουμε τη νέα συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Αζερβαϊτζάν, θα είναι σημαντικό να επιβεβαιώσουμε τη δέσμευσή μα και την αιμονή μα στην αιρεσιμότητα σε ό,τι αφορά τι συνθήκε αυτέ ε, για την ε, σύνδεση και σε ό,τι αφορά το σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θεμελιωδών δικαιωμάτων, κράτο δικαίου, δημοκρατία. Όλα αυτά θα πρέπει να αποτελούν πυρήνα των συμφωνιών. Δεν μπορούμε να τα παραβλέπουμε και αυτό θα πρέπει να το εξετάσει το Κοινοβούλιο και να το εξετάσει διαρκώ και σε μετέπειτα χρονική στιγμή. Εν τω μεταξύ, λοιπόν, μια και οι εκπρόσωποι τέτοιων ανθρώπινων δικαιωμάτων ε, φυλακίζονται και εκφοβίζονται, θέλουμε η ύπατη εκπρόσωπο, η κυρία Μογκερίνη, να καταπιέσει, να καταδικάσει, συγγνώμη, τις ε, παραβιάσεις αυτές στο Αζερβαϊτζάν με του πιο καυστικού όρου και να ζητήσει επίση και αυτή απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, και η Πρόεδρο. Η κυρία Γκόμα έχει τώρα το λόγο για δύο λεπτά. Όταν μιλάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για το κράτο δικαίου, ότι αποτελούν τη βάση των δράσεών μας ε, κατά των τρίτων χωρών μέσω των συμφωνιών που έχουμε διαπραγματευτεί με αυτές που είναι υποδιαπραγμάτευση στην περίπτωση του Αζερβαϊτζάν. Όλα αυτά δεν είναι ρητορικά. Μιλάμε προκειμένου άνθρωποι σαν και εσά, ε, κυρία Μάλμστρομ, όπω και η κυρία Μογκερίνη, πραγματικά να ε, πετύχουν, να ισχύουν όλα αυτά. Δεν είναι όλα αυτά κατ' κατ όνομα μόνο. Και αυτό που συμβαίνει στο Αζερβαϊτζάν είναι σκανδαλώδε. Και αυτό φαίνεται και στην υπόθεση του Μεχμάν Χουζαϊνόφ, αλλά η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσαμε να αναφέρει πάρα πολλού τέτοιου ακτιβιστέ, ε, όπω την κυρία Σμαϊλαβά, τον Γκουγκαρ Μέρφοφ. Ε, τον κύριο Μοχτάρη, ο οποίος ε, απήχθη στη Γεωργία και μεταβιβάστηκε στην Αζερβαϊτζάν να φυλακιστεί και να μασανιστεί. Γιατί, γιατί αυτοί οι γενναίοι άνθρωποι βγήκαν να εκθέσουν τη διαφθορά που μαστίζει αυτό το καθεστώς, ε, Αλιεφ. Πραγματικά είναι φρικτό το γεγονός ότι παρά όλες αυτές τις αρχές, τελικά ο κόσμος αυτό ο οποίο κάνει τι διαπραγματεύσει και πρότεινε στο κοινοβούλιο να δώσει τη συνένεσή του, τελικά κάνουν το αντίθετο. Είναι όνειδο. Εμεί περιμένουμε ότι θα δράσετε βάσει των αρχών αυτών και θα πρέπει να γίνει κάποια αξιολόγηση τη κατάσταση. Η κατάσταση είναι αυτή που περιέγραψαν οι συνάδελφοι, που πήραν τον λόγο προηγουμένω στην περίπτωση του Μεχμάν Χουσέινοφ. Φαίνεται σαφέστατα το επίπεδο της καταποίησης των βασανιστήριων που υπόκειται οι άνθρωποι αυτοί. Την εβδομάδα αυτή ένας από του αδέλφους μας, ο κύριος Νικολάη, μας μοίρασε μια επιστολή που συνέταξε, αναγκάστηκε να συντάξει. Γιατί αν διαβάσετε την επιστολή αυτή μου θυμίζει τις επιστολές που έστελναν οι άνθρωποι υπό την δικτατορία του Σαλαζάρ στην δική μου χώρα και υπό την δικτατορία του Τσαουσέσκο για να υποκριθούν ότι τάχα υπό συνθήκες εξαιρετικές, ε, εξαιρετικά άσχημες, αλλά πήγαιναν καλά για να εγκρίνουμε το ψήφισμα που θα εγκρίνουμε σήμερα. Και επίση κάτι πολύ σημαντικό που ανέφερε ο συνάδελφο Ουρμπαν Κρέσπο, η διαφθορά η οποία υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Αζερβαϊτζάν καταδεικνύει ότι ακόμα και εδώ στο Κοινοβούλιο, όπως ήταν το 2013, στις εκλογές στο Αζερβαϊτζάν, υποστηρίζονται ουσιαστικά δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό. Το θέμα δεν είναι μόνο το Αζερβάιτζαν. Το θέμα δεν είναι μόνο να υποστηρίξουμε την καταπολέμηση τη διαφθορά και την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Το θέμα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, η κυρία Ζόφκο, Ζηλιάνα. Παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις ε, συζητήσεις που είχαμε ε, για το Μεχμάν Χουσεϊνοφ, διότι την χάνω σκιώδη εισηγήτρια του ΕΛΚ για το Ζερβαϊτζάν και διαπραγματεύτρια της ομάδας μου για το συγκεκριμένο ψήφισμα. Πραγματικά είναι σημαντικές οι διμερείς μας σχέσεις με το Αζερβαϊτζάν και θα πρέπει να δώσουμε προσοχή στη νέα εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Αυτό θα πρέπει να είναι στον πυρήνα της συζήτησης αυτής. Ο, Μεχμάν Χουσεϊνόφ είναι ένας blogger κατά της διαφθοράς και έχει καταδικαστεί σε διετή φυλάκιση. Επειδή κατήγγειλε στη συνέχεια ε, δημόσια ε, την κακομεταχείριση του και τους βασανισμούς του από την αστυνομία και κατήγγειλε και άλλα κακό κείμενα δύο μήνες πριν αφαιθεί ελεύθερος, πριν αποφυλακιστεί για τη λίγη ποινή του ε, θέλουν να την παρατείνουν κατά 5 ή 7 έτη. Το ψήφισμα ζητεί να αφαιθεί άμεσα ελεύθερος και να του παρασχεθεί ιατρική βοήθεια θα πρέπει να στείλουμε το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προτίθεται ε, να διακόψει τις σχέσεις με το Αζερβαϊτζάν, αλλά ότι ε, υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις στη συνεργασία αυτή. Θέλουμε μεν να συνεργαζόμαστε, αλλά με συγκεκριμένες βάσεις. Και μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εκείνη που μπορεί να βοηθήσει τη χώρα για να ενισχυθούν τα δικαιώματα και το κράτο δικαίου. Απευθύνω έκκληση λοιπόν να φεθούν ελεύθεροι όλοι οι κρατούμενοι συνείδησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τηρεί ε, τις αρχές της και απέναντι σε όλες τι χώρε με τι οποίε συνεργάζεται. Όχι μόνο για το Ζερβαϊτζάν και ε, τις τρεις χώρες της περιοχής. Αυτά δεν μπορούμε να τα απεμπολούμε και ούτε να είμαστε επιλεκτικοί στην αντιμετώπιση μιας χώρας. Είναι καλό το ψήφισμα λοιπόν γιατί προειδοποιεί το Αζερβαϊτζάν. Ακούσαμε για τη διαφθορά από 180 χώρες, είναι στη θέση 163, είναι τραγικά αυτά τα πράγματα. Χρησιμοποιούν τα κονδύλια για να αγοράζουν επιρροή ε, ασκούν πιέσει και εξαγοράζουν κανονικά δημοσιογράφου. Ε, μας ανησυχούν αυτέ οι πρακτικέ, θα πρέπει να τερματιστούν και ελπίζω να αφαιθεί ελεύθερο ο Χουσέινοφ και να έχει ιατρική περίθαλψη. Θα πρέπει να αφαιθούν ελεύθεροι όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι, όλοι οι κρατούμενοι συνείδησης, διότι είναι απαράδεκτα πράγματα στον 21ο αιώνα αυτά η συνεργασία μας με τις χώρες που είναι εταίροι μας θα πρέπει να βασίζεται σε αμοιβέ αρχές και αξίες. Και μία από αυτές είναι η ελευθερία της έκφρασης. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αυτά τα πράγματα δεν χωράνε παζάρια και εκπτώσεις. Είναι τα θεμέλια της συνεργασίας μας και των σχέσεών μας με τις τρίτες χώρες, ανεξαρτήτως περιοχής ή πλούτου που έχουν. Γι' αυτό θα αγωνίζομαι ε, όσο είμαι βουλευτή. Ο κύριο Στέτιν, αν 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι. Καλό για την άμεση απελευθέρωση και του κυρίου Χουσμάν, ε, ο οποίο έχει φυλακιστεί στο Αζερβαϊτζάν γιατί προσπάθησε να διαμαρτυρηθεί κατά τη διαφθορά και τη αδικία. Υπάρχουν και άλλοι πολιτικοί κρατούμενοι μα στο Αζερβαϊτζάν, δεν είναι ο μόνο ο κύριος Αφκάν Μουχτάρλη, ο οποίος απήχθη ε, γιατί αποκάλυψε το τι κάνουν οι μυστικές υπηρεσίες στη Γεωργία. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα συστήματα δίωξης ε, εξάγονται και σε άλλες χώρες. Η απαγωγή που σας ανέφερα έγινε σε άλλη χώρα από το καθεστώς του Αζερβαϊτζάν. Πολλές φορές λένε και κατηγορούν μάλλον την Ιντερπόλ ότι δεν ε, ε, εκδίδει αυτούς που έχουν διαφωνήσει με το καθεστώς και την κυβέρνηση. Η Ιντερπόλ πολλές φορές προφανώς δεν μπορεί να εκδώσει πολιτικούς ε, αντιπάλους και κρατουμένους. Είναι κατά των αρχών μας και το ίδιο του άρθρο 3 του εσωτερικού της κανονισμού. Η Ιντερπόλ δεν παίρνει μέρος σε εσωτερικές υποθέσεις των διαφόρων χωρών με πολιτικό μάλιστα περιεχόμενο η Ιντερπολ αρνήθηκε και την σύλληψη τριών βουλευτών όπως είχε ζητηθεί από τον Πακού ε, για να προσπιστεί την ελευθερία της σκέψης, της έκφρασης και των ε, πολιτικών ε, φρονημάτων στο Αζερπαϊτζάν. Εδώ πρέπει να ασχοληθούμε σφαιρικά με το θέμα του Αζερπαϊτζάν. Κυρία Πόστ, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα σας, Επίτροπε και συνάδελφοι. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τρίτο ψήφισμα για το Αζερβαϊτζάν και τι παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια τη θητεία μα. Είναι η στιγμή η κυβέρνηση τη χώρα να λάβει σοβαρά υπόψη τι εκκλήσει μα. Ζητούμε την άμεση και ανεφόρον απελευθέρωση του κυρίου Χουσέινοφ και όλων των άλλων πολιτικών κρατουμένων, δικηγόρων, ακτιβιστών, πολιτικών αντιπάλων, ε, ακτιβιστών κατά τη διαφορά, ανεξάρτητων δημοσιογράφων και μπλόγκερ στο Αζερβαϊτζάν. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν συλληφθεί και βασανίζονται στη φυλακή διότι ασκούν την ελευθερία της έκφρασης και επειδή επικρίνουν την κυβέρνησή τους. Αυτό δεν είναι έγκλημα. Οι ε, αξιωματούχοι ε, της χώρας πρέπει να καταλάβουν ότι αποτελεί δικαίωμα. Κάποιοι από αυτοί ε, εκτίουν ποινές δεκαετίας, καθήλξης διότι απλώς διαμαρτυρήθηκαν κατά της διαφθοράς της κυβέρνησής τους. Όμως η ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και του τύπου προφανώς καταπιέζεται και καταπατάται στο Αζερβαϊτζάν. Δεν μπορούμε να δεχτούμε την καταπίεση των ε, ΛΟΑΔ, των ε, δημοσιογράφων και ανεξάρτητων δημοσιογράφων, των blogger και όσων θέλουν να εκφραστούν ελεύθερα. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προβλέψει κυρώσει κατά της τάση αυτής των ε, κυβερνώντων στο Αζερβαϊτζάν. Θα πρέπει να ανασταλεί οποιαδήποτε χρηματοδότηση για τις κρατικέ δομέ επιχειρήσει και κοινέ επιχειρήσει στο Αζερβαϊτζάν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίτροπε. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Καρίν. Κύριε, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ω πρόεδρο τη αντιπροσωπεία για τι σχέσει με τι χώρε του Νοτιού Καυκάσου, πρέπει να πω ότι έχουμε δει μια σοβαρή ε, καμπή στι σχέσει μα με το Αζερβαϊτζάν. Μήνα με το μήνα και χρόνο με το χρόνο, η πρόοδο που έχει γίνει, ώστε να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει μια ισχυρή σχέση συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Αζερβαϊτζάν, είναι μια πρόοδο που μπορούμε να την δούμε με άλματα ε, και βήματα. Ω πρωταθλήτρια των δημοκρατικών, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη ελευθερία του λόγου και τη έκφραση ανά τον κόσμο, δεν θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραβλέπει την ε, καταπίεση και δίωξη οποιαδήποτε άτομα από οποιαδήποτε κυβέρνηση. Ακόμη και αν είναι μεγάλη πρόοδο που έχει γίνει στι διεθνεί μα συμφωνίε, ε, δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε τα άτομα και τι ατομικέ του ελευθερίε. Από αυτέ οι αυτοί πρέπει να θεωρηθούν πρώτοι. Στο ψήφισμα λοιπόν που έχουμε μπροστά μα σήμερα υπάρχουν πολλά τέτοια στοιχεία. Το κοινοβούλιο μα πρέπει να ενισχύσει το μήνυμα του, καλώντα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και την κυβέρνηση του Αζερβαϊτζάν ώστε να πιέσουν ε, ε, να υπάρξει προστασία για όσους κατηγορούνται, να τους παρασχεθεί ιατρική περίθαλψη, πρόσβαση σε συνήγορο, ε, ε, δικαίωμα επίσκεψης από τις οικογένειές τους και τα μέλη των οικογενειών τους για όσους κατηγορούνται άδικα. Οι καλές σχέσεις που έχουμε οικοδομήσει με κόπο μέσα από τα χρόνια με το Αζερβαϊτζάν έχουν αποδώσει καρπού. Θα πρέπει να, να καλέσουμε μάλλον ε, θα πρέπει να πούμε ότι και το δικαίωμα επίσκεψη στον κύριο Χουσέινοφ, ε, εφόσον γίνει δεκτό, θα ήταν ένα πολύ καλό βήμα για την επίλυση του όλου προβλήματο. Οι σχέσει μα θα πρέπει πάντοτε να αντικατοπτρίζουν τι αξίε μα. Όμω παρομοίω θα πρέπει να σεβόμαστε και όλου του εταίρου μα. Ευχαριστώ. Ε, δυόμιση λεπτά, κυρία Νικολάη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ως εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Αζερβαϊτζάν, θα ήθελα να πω το εξής. Τρία ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης για το Αζερβαϊτζάν έχει εξελιχθεί ε, θετικά και προετοιμάζουμε αυτόν τον καιρό μια συμφωνία εταιρικής σχέσης. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να κάνουμε μια πάρα πολύ σοβαρή συζήτηση ε, για ε, το τι επιπτώσεις έχουν οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για μια τρίτη χώρα. Εμείς όλοι είμαστε καλόπιστοι και προσπαθούμε να έχουμε επικοδομητικό διάλογο με τις ε, αρχές της χώρας αυτής, με τις κρατικές αρχές. Θυμηθείτε και τις επιτυχίες που είχαμε στα ανθρώπινα δικαιώματα. Την περίπτωση του κυρίου Ντομάτοφ και προσπαθούμε να λύνουμε ε, τα προβλήματα με έναν τρόπο σωστό, αξιοπρεπή και όχι συγκρουσιακό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ε, αναπτύσσει και μια διπλωματία και ε, στα πλαίσια ενός μονίμου διαλόγου. Έτσι έχουν αφαιθεί ελεύθεροι 146 πολίτες και είναι πολύ θετικό αυτό. Κοιτάξαμε πολύ προσεκτικά αυτές τις αιτιάσεις και την κατάσταση ε, και άλλων. Στο μεταξύ, μου έχουν δοθεί κάποιες εξηγήσει από τις αρμοδίες αρχές και τις διοικητικές και μου είπαν ότι επιτέθηκε σε ένα δεσμοφύλακα ε, και μάλιστα με δόλο. Ο κύριος Χουσέινοφ κάνει απεργία πείνας και έμαθα και μάλιστα το επιβεβαίωσα κιόλα. Συνάδελφοι, όταν ε, συντάσσουμε ένα ψήφισμα που έχει να κάνει με ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλά θα κάνουμε πρώτα απ' όλα να γνωρίζουμε τα πραγματικά περιστατικά, να ακούμε όλες τις πλευρές, να είναι πολύ τεκμηριωμένη αυτή η πρόταση, ε, να μην είμαστε μεροληπτικοί υπέρ της μίας πλευράς ή της άλλης, γιατί μπορεί να ε, μας λείπουν στοιχεία. Πάντα κινδυνεύουμε από παραπληροφόρηση, από ψευδείς ειδήσει, fake news κτλ. Και αυτό θα επηρεάσει και τη διπλωματική μας δράση. Δύο λεπτά, κυρία Χάουτα. Α, συγγνώμη. Δέχεστε μια γαλάζια κάρτα από την Άννα ε, Κυρία Νικολάη, θα συμφωνήσετε ότι είναι τελείως απαράδεκτο το καθεστώς του Αζερβαϊτζάν να εξαγοράζει Ευρωπαίους πολιτικούς, όπως είναι ο κύριος Πέντρο Αγκραμόντ, που είναι αυτή τη στιγμή γερουσιαστή στην Ισπανία χωρίς να έχει διερευνηθεί καθόλου αυτή η περίπτωση διαφθοράς συμφωνείτε ότι αυτό προκαλεί τεράστια ε, ε, ζημιά στην αξιοπιστία των ευρωπαίων πολιτικών και της ευρωπαϊκής δράσης. Εάν δωροδοκούνται και εξαγοράζονται από ένα τέτοιο καθεστώς ευρωπαίοι πολιτικοί, όπως είναι το καθεστώς του Προέδρου Αλίεφ. Απάντησε. Κυρία Νικολάη, ευχαριστώ Ανά. Συμφωνώ απολύτω μαζί σου. Δεν την ήξερα εγώ αυτή την περίπτωση του Ισπανού πολιτικού. Πρώτη φορά την ακούω. Ελπίζω να ε, διευκρινιστεί και να διαλευκανθεί και ελπίζω να μην είναι μια απλή κατηγορία και ε, ένας ισχυρισμό εναντίον ενός πολιτικού, γιατί ούτε αυτό θα ήταν ε, παράδεκτο. όταν κάνουμε ψηφίσματα θα πρέπει να βλέπουμε και τα θετικά. Να μην γίνονται καταχρήσεις, να μην φυλακίζονται οι πολίτες, συμφωνώ. Αλλά εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να κάνουμε κάτι χειροπιαστό αυτό για τους πολίτες. Ο κύριος Καστάλντο, ένα λεπτό. sorry. συγγνώμη, η κυρία Χάουταλα προηγουμένω. Δύο λεπτά. Πρόεδρε, το υπερήφανο και σημαντικό αυτό έθνος του Νοτιού Καυκάσου ε, γιόρτασε τα 100 χρόνια ανεξαρτησίας του πριν από ένα χρόνο περίπου. Και τι έγινε. Στο περιθώριο της τελετής αυτής, τέσσερι ε, τέσσερα μέλη του ανεξάρτητου συνασπισμού ε, συνελήφθησαν. Είναι αυτό δημοκρατία. Είναι δημοκρατία που θεμελιώθηκε σε πραγματικές αρχές δημοκρατίας και θέλει να γίνει πρωταγωνιστής στη διεθνή κοινότητα και να έχει στενότερους δορισμού με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η χώρα που ως δημοκρατικό καθεστώς πρέπει να προστατεύει τις ελευθερίες και τα δικαιώματα των πολιτών της. Δεν μου φαίνεται να είναι έτσι. Και έχω σημαντική σχέση και ιδιαίτερη σχέση με τη χώρα αυτή, γιατί η γιαγιά μου γεννήθηκε στον Πακού. Το 1916 έγινε 100 και έχει ακόμα να πει υπέροχε ιστορίε για την παιδική τη ηλικία και το τι έζησε στο Αζερβαϊτζάν. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε ότι ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να ενισχύσει τι συμβασιακέ τη σχέσει με το Αζερβαϊτζάν, η χώρα αυτή δυστυχώ ε, αποτρέφεται των διεθνών τη υποχρεώσεων στο Συμβούλιο τη Ευρώπη, στον ΟΣΑ, στον ΟΑΣΕ μάλλον, και δεν λαμβάνει υπόψη την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης και τους εκπροσώπους των, της των μέσων μαζική Ενημέρωση των ΑΣΕ που ανησυχούν πολύ για την κατάσταση στη χώρα και ιδίω για την κατάσταση υγεία του κυρίου Χουσίνοφ. Εμεί, ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να απευθύνουμε έκκληση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΕΔ να κάνουν ό,τι περισσότερο μπορούν Διότι αν η κυβέρνηση του Αζερβαϊτζάν θέλει στενότερε σχέσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να ε, απελευθερώσουν ανεφόρον αμέσω του πολιτικού κρατουμένου και βεβαίω και τον κύριο Μεχμάν Χουσέινοφ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Καστάλντο δεν είναι εδώ. Εάν έρθει θα λάβει το λόγο. Ο κύριος Κολομπιέ για δυόμιση λεπτά. Πρόεδρε, Στι ε, ε, συνεδριάσει μα στι μας, στις μας του Πέμπτη το πρωί που γίνονται για λόγου καλή συνείδηση, μιλάμε για την περίπτωση του Μεχμάν Χουσέινοφ τώρα, ε, για τη διετή του ποινή, επειδή κατήγγειλε το καθεστώ του Αλίεφ. Ναι, είναι αποτελεσματικό αυτό το καθεστώ. Όμω τι έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την κυβέρνηση αυτή. Να θυμίσω ότι στι 16 Νοεμβρίου του 2016 το Συμβούλιο ανέθεσε στην Επιτροπή Εντολή για να ξεκινήσει μια σφαιρική συμφωνία με το Αζερβαϊτζάν και τι σχετικέ διαπραγματεύσει. Στι 7 Φεβρουαρίου του 2017 οι διαπραγματεύσει αυτέ ξεκίνησαν μετά την επίσκεψη του Προέδρου Αλεύ στι ε, Βρυξέλλε και τι 11 Ιανουαρίου 2018 εγκρίθηκαν νέε προτεραιότητε για την εταιρική σχέση. Προβλέπεται ιδίω να είναι πιο ευέλικτο το καθεστώ των θεωρήσεων, το σύστημα των θεωρήσεων. Ξέρουμε ότι έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια αιμονή να φέρει ε, άλλα κράτη και έθνη σε μια εποχή ψυχρού πολέμου πάλι με τη Ρωσία. Εδώ αυτή η αποκαιοκρατική μας πολιτική θέλει και θα οδηγήσει ε, και σε ε, συντρούσει στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Θα πρέπει να επιδιώξουμε, πολύ το είπατε, στενότερες σχέσεις με το καθεστώς του Μπακού. Όμως αυτή τη στιγμή Υπάρχει μια ολόκληρη σχέση που χτίζεται μεταξύ του Αζερβαϊτζάν και των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ε, εξασφάλιση της τροποδοσίας μας σε ε, κάψιμα θα πρέπει να περάσουμε και από τη Ρωσία με τους αγωγούς ε, αερίου που χτίζονται. Θα πρέπει λοιπόν η συνάδελφο Νικολάη, ε, η συγγήτρια τη έκθεση του Κοινοβουλίου για αυτή τη νέα συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Αζερβαϊτζάν, να σκεφτεί σοβαρά και αυτή τη διάσταση. Αν δω τι λέει η Γαλλική Εφημερίδα Λιμπερασιών ε, και για παρόμοια υπόθεση παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπήρξε καταπίεση τη ελευθερωτυπία του Γιουνί ε, Σάχαροφ στο Αζερβαϊτζάν στο πρακτορείο τύπου της χώρας ε, καταγέλθηκε ε, η συμπεριφορά του, ενώ πρόκειται για ένα όργανο ουσιαστικά της κυβέρνησης, ε, όταν μιλάμε για αυτό το πρακτορείο τύπου. Ε, η Άλντε τι έχει να πει για το μαρτύριο που περνάει ο λαός της Αρμενίας στο Ναγκόνο Καραμπάχ ε, στο ε, εξαιτία του και τη κυβέρνηση του Μπακού. Ε, τα θύματα τη κατάσταση στο Νότιο Κάφκασο είναι ο λαό τη Αρμενία. Σταματήστε λοιπόν αυτέ τι κινήσει ξεπλήματο τη συνείδησή σα και σταματήστε τη σχέση σα με το καθεστώ του Μπακού. Ευχαριστούμε κύριο Σόγκορ η παραβιάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποφασίζουν μια λυπηρή πραγματικότητα στο Αζερβαϊτζάν και σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία έχουμε πάνω από 100 πολιτικού ε, κρατούμενου στο Νότιο Κάφκασο, στην χώρα του Ναυτικού Καυκάσου, όπου το καθεστώ επίση ε, ελέγχει στενά τα μέσα ενημέρωση. Σύμφωνα με τον αδερφό του φυλακισμένου blogger και ακτιβιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο οποίο βρίσκεται σε απεργία πείνα, όλοι οι γνωστοί προασπιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογράφοι περνούν τουλάχιστον κάνα δύο χρόνια στη φυλακή. Και αυτή η πρακτική επιδεινώνεται από μια κοινή πρακτική, όπου οι αρχέ τη Αζερβαϊτζάν απαγγέλουν όλο και νέε κατηγορίε κατά των πολιτικών κρατουμένων και δεν τελειώνουν τελικά ποτέ αυτέ οι ε, φυλακίσει. Ξέρουμε ότι πρόκειται για την πέμπτη αυτή περίπτωση του τελευταίου μήνε. Το Αζερβαϊτζάν λοιπόν συχνά ε, και εδώ και καιρό προσπαθεί να προστατευτεί από το κριτική της των δυτικών κρατών, χρησιμοποιώντας τη στρατηγική θέση που έχει και την περιφερειακή συμμαχία στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας, καθώς και το γεγονός ότι είναι σημαντική η χώρα για την Ευρώπη για την ε, μείωση της εξάρτησης από το ρωσικό αέριο. Αλλά Επίση είναι γνωστό για τη χρήση ε, δωροδοκία και ε, ξένων ταξιδιών για του ε, αξιωματούχου τη Δύση. για να απαλύνει την κριτική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δώσει λοιπόν ένα σαφέ μήνυμα ότι παίρνει στα σοβαρά όλε αυτέ τι παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι βάζει τα θέματα αυτά στο επίκεντρο της νέας αυτή συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση και Αζερβαϊτζάν. Στην φάση αυτή είναι σημαντικό να ζητήσουμε άμεση και αναφορών απελευθέρωση του κ. Χουσέινοφ από τις αρχές της το Αζερβαϊτζάν και να σταματήσουν ε, οι κατηγορίες, ε, να αρθούν οι κατηγορίες ε, κατά αυτού. Επίσης, άμεση και ανεφόρον απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων, δημοσιογράφων, ακτιβιστών των ανθρώπινων δικαιωμάτων και άλλων ακτιβιστών για την κοινωνία των πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Κραπίνη έχει τώρα το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Ευθύς εξ αρχής θα ήθελα να πω ότι πρόκειται για ένα απαραίτητο ψήφισμα και θα πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή στην κυβέρνηση του Αζερβαϊτζάν για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ωστόσο, είναι σημαντικό να μιλήσουμε και για την εξαγωγή διαλόγου με το Αζερβαϊτζάν, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τι παραβιάσει αυτών αλλά και την καταπολέμηση της δημοκρατίας στην περιφερειακή σταθερότητα, τη χειραγώγηση που θα πρέπει φυσικά να καταπολεμήσουμε. Σε ό,τι αφορά δε τις δημοκρατικές αρχές, το Ζερβαϊτζάν έχει προσυπογράψει στις σχετικές αρχές του Συμβουλίου της Ευρώπης και πλέον διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν ανησυχίες σε ό,τι αφορά και τις διεθνείς οργανώσεις και τα μέσα ενημέρωσης. Οι Ευρωπαίοι λοιπόν έχουν καθήκον να τα εξετάσουν όλα αυτά και θα πρέπει να αναπτύξουμε λοιπόν αυτή την εταιρική σχέση με τις χώρες ε, της Ανατολικής Γειτονίας. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να κατανοήσουν και οι χώρες αυτές τη σημασία των ψηφισμάτων όπως το σημερινό ψήφισμα, το οποίο είναι θεωρώ ισορροπημένο. Το ψηφίσμα αναφέρει τα θετικά στοιχεία για την απελευθέρωση, για παράδειγμα, ακτιβιστών, δημοσιογράφων. Και θεωρώ ότι η οδός που θα πρέπει να ακολουθήσει, αν θέλετε, στο μέλλον του Αζερβαϊτζάν, θα πρέπει να οδηγήσει προς την Ευρώπη. Θα θέλαμε λοιπόν να τονίσουμε ότι το κράτος είναι αυτό που επικρίνουμε, όχι τους πολίτες. Το κράτος ευθύνεται για τις παρεμβάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα πρέπει να συνεργαστούμε με τον Πακού και να συζητήσουμε ακριβώ τα θέματα αυτά. Πιστεύω λοιπόν ότι η συμφωνία του Αζερβαϊτζάν που ξεκίνησε το 1997 θα πρέπει να συνεχίσει. Ευχαριστώ. Ε, ο κ. Ντέμε Μάκερ. Ε, πρόεδρε και ε, Επίτροπε, δεν συμφωνώ με κάποιου συναδέλφου που προσπαθούν να σχετικοποιήσουν ή να οροποιήσουν την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων με το επιχείρημα ότι έχει γίνει και πρόοδοι. Κοιτάξτε, έχει καταστεί παγκόσμιο προμηθευτή τη αυλή στην καταδίωξη των blogger. Αυτό είναι εξαγωγικό προϊόν, όχι πολύ ζηλευτό, αλλά σκοτίστηκε τώρα ο πρόεδρο Αλίεφ. 150 πολιτικοί αντίπαλοι και δημοσιογράφοι περίπου είναι φυλακοί. Και σήμερα καλούμε να αφαιθεί ελεύθερο ένα νέο ακτιβιστή, ο Μεχμάν Χουσεϊνοφ, που έχει μια κριτική πένα και έχει βάλει ένα καθρέφτη αντιμέτωπο με το καθεστώς ε, και αυτός ο καθρέφτης δεν δείχνει καθόλου ωραία εικόνα γιατί ε, ο λαός ε, στενάζει με τη φτώχεια και η πολιτική ελίτ γύρω από τον πρόεδρο Αλίεφ γιορτάζει και είναι πολύ ψηλό το τίμημα που πληρώνει ο κύριος ε, Χουσέινοφ. Ε, με κατασκευασμένες κατηγορίες έχει φυλακιστεί για δύο χρόνια. Το Μάρτιο κανονικά αποφυλακίζεται και τώρα ευαπηλείται με νέες κατηγορίες και φυλάκιση και κάθερξη μέχρι 7 έτη. Ε, καλό είναι να ενισχυθεί η σχέση μας με το Αζερβαϊτζάν, αλλά χωρίς να παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα θεμελιώδη, η ελευθεροτυπία κτλ. Η κυρία Πάρκερ για 2,5 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ένας ελεύθερος ε, ε, τύπος ε, που να ανθεί είναι προϋπόθεση για μια δημοκρατία. Όταν αυτό δεν ισχύει, αυξάνεται η απόσταση ανάμεσα στο λαό και τους πολιτικούς που τον εκπροσωπούν. Είναι μεγάλη διαφθορά, δυστυχώς, στο Αζερπαϊτζάν. Είπαμε ότι είναι στη θέση 163 ε, από το δίκτυ ελευθεροτυπίας από 180 χώρες. Ο ε, Μεχμέτ Χουσέινοφ είναι η ενσάρκωση εκείνων που προσπαθούν να καταγγέλουν τα προβλήματα της διαφθοράς ε, στο Αζερπαϊτζάν και τι κάνει αυτό στο λαό πολυτελείς κατοικίε και άλλα αγοράζουν Όλα αυτά τα έχει καταγγείλει και οι δημοσιογράφοι χωρί σύνορα καταγγέλουν ότι μπορεί να πεθάνει και στη φυλακή γιατί κάνει απεργία πείνα. Πολλοί ε, είναι εκείνοι που έχουν αρχίσει και αυτοί απεργία πείνα και έχει έρθει η ώρα πολιτική πολιτικοί να ακούσουν το λαό και να αρχίζουν να διορθώνουν τα κακό σκήμενα τη δημοκρατία και να επιτρέψουν να αναπτυχθεί μια ε, ε, γνήσια δημοσιογραφία και ελευθεροτυπία πραγματική σε αυτό το τόπο. Ο κύριος Κέλλη για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ καταδικάζω ότι η κατάσταση στο Αζερβαϊτζάν γιατί παραβιάζει η κυβέρνηση τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθεροτυπία κτλ. Ε, φημώνεται ε, όποιος ε, καταγγέλει και κατηγορεί την κυβέρνηση δημοσιογράφοι και bloggers βλέπουν να τους απεγγέλλονται νέες κατηγορίες όταν τελειώνει η ποινή τους για να παραταθεί. Η συμμετοχή του Αζερβαϊτζάν στην εταιρική σχέση με την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ανατολική Γειτονία, σημαίνει ότι έχει δεσμευτεί ε, σε κάποια πράγματα και στο Συμβουλίο της Ευρώπης. Αλλά αυτά τα υπονομεύουν οι αρχές. Γι' αυτό καλό την κυβέρνηση του Αζερβαϊτζάν να ανταποκριθεί στις διεθνείς υποχρεώσεις και να υλοποιήσει και να σεβαστεί τι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Να αφήσει ελεύθερου όσοι αδίκως κρατούνται, ιδιαίτερα τον κύριο Χουσέινοφ, τον οποίο αναφέρθηκαν και άλλοι ομιλητές, και κάνει απεργία πείνα από το Δεκέμβριο του 2018 διαμαρτυρία. Είναι επιλεκτικέ οι διώκτησει και θα πρέπει να τερματιστεί αυτή η πρακτική. Φυσικά θα πρέπει να επιτρέπεται να επικρίνει κάποιο την κυβέρνηση. Δεν χωράνε τέτοια μέτρα σε μια χώρα που έχει δεσμευτεί υπέρ του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και της προστασίας των ανθρωπινών δικαιωμάτων και θέλει να έχει και στενές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ε, η κυρία Τζούλι Γουόρτ, παρακαλώ για δύο λεπτά. The EU's... Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ζερβαϊτζάν Πρέπει να είναι πολύ πιο αυστηρή. Η κοινωνία των πολιτών ε, προσπαθεί να αναπτυχθεί σε εχθρικό περιβάλλον. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσει αναγκάζονται να ε, κλείσουν. Και ε, όσοι προσπαθούν να εκφράσουν μια διαφορετική άποψη εξορίζονται ή φυλακίζονται. Ο Μέχμαν βρίσκεται τώρα στην 130η περίπου μέρα τη απεργία πείνα του. Έχει υποστεί βασανιστήρια πολλέ φορέ και η κατάσταση είναι πολύ επικίνδυνη. Του προηγούμενου μήνε υπήρξε ανησυχητική αύξηση στον αριθμό απεργιών πείνα ε, στον κόσμο. Η Λέιλι Κούβαν στο Κουρδιστάν, και ο κύριος Ράκλεφ ε, και ο κύριος Μαχάμιτ στο Ιράν. Όλοι αναγκάστηκαν να καταφύγουν στην απεργία πείνας ε, σε κατάσταση απελπισίας. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτές τις δημόσιες, ε, αυτές τις καταστάσεις μάλλον και να κάνουμε δημόσιες δηλώσεις απαιτώντας από την κυβέρνηση του Αζερβαϊτζάν να απελευθερώσει αμέσως και ανεφορών τον Μέιγμαν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγορεί και πονηδίζει κάθε χώρα που παραβιάζει τα ανθρώπινα και δημοκρατικά δικαιώματα ασχέτως των οικονομικών δεσμών που έχει μαζί του. Ε, θα πρέπει να αναλυφθεί και δράση. Καλό την Ευρωπαϊκή λοιπόν, Ένωση και τα κράτη-μέλη να επιβάλλουν κυρώσει. Κυρώσει όχι μόνο στον πρόεδρο, αλλά και κατά των υπουργών του. Διότι ω τώρα δεν έχουν στοχευθεί. Ευχαριστούμε και τώρα περνάμε στη διαδικασία Κατσδιάη. Ο κύριος Φαρία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε. Ο Μεχμάν Χουσέινοφ, blogger και δημοσιογράφο, ε, υπεύθυνο του Ινστιτούτου για την Ελευθερία και την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων, η ΑΕΡΕΦΕΣ, εκτύπηνε φυλάξει δύο ετών. Ε, δεν είναι μεμονωμένη η περίπτωση αυτή. Οι αρχέ του Αζερβαϊτζάν και η κυβέρνηση τη χώρα έχουν ε, πραγματικά εμποδίσει του δημοσιογράφου και ακτιβιστέ που θέλουν να καταγγείλουν τη διαφορά στη χώρα με διώξει, αυθαίρετε συλλήψει και άδικε καταδίκες. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που περνάμε ψήφισμα για το Αζερβαϊτζάν στο σώμα αυτό. Πιστεύω ότι ήρθε η στιγμή να πούμε φτάνει, ω εδώ και μη παρέκει. Δεν ε, μπορούμε παρά να απαιτήσουμε από την κυβέρνηση του Αζερβαϊτζάν να πάψει τη δίωξη των πολιτών, τη κοινωνία των πολιτών, ε, να αφήσουν του δημοσιογράφου να εκφράζονται ελεύθερο στη χώρα και να απελευθερώσουν αμέσω τον κύριο Χωσέινοφ και όλου του άλλου πολιτικού κρατουμένου και ακτιβιστέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να τηρήσει μια ξεκάθαρη στάση βάσει τη ε, αρχή τη ελευθερία ε, του λόγου και τη ελευθεροτυπία, κάτι που βρίσκεται στην καρδιά των θεμελιών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, κυρία Επίτροπε, δεν είναι αντάλλαγμα σε διαπραγματεύσει, ούτε μπορούν να γίνουν κάτι τέτοιο. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει την ευθύνη αναστολή τη χρηματοδότηση προ την ε, κυβέρνηση του Αζερβαϊτζάν που δίνεται υπό τη μορφή βοήθεια. Ευχαριστούμε κύριο Πόσπισιλ. Ευχαριστώ. Επίτροπε, Ευχαριστώ γιατί θα ήθελα να συμφωνήσω με όλους τους συναδέλφους που ζήτησαν να τηρήσουμε εδώ μια αυστηρή στάση ε, απέναντι στο Αζερβαϊτζάν για την περίπτωση του κυρίου Χουσέινοφ. Εγώ είμαι πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης και πιστεύω ότι θα πρέπει να επικρίνουμε το Αζερβαϊτζάν και να είμαστε αυτοί μαζί του και σε άλλε περιπτώσει παραβίαση του κράτου δικαίου. Το 2017 έγινε μεταρρύθμιση, α πούμε, του δικαστικού συστήματο, τη εργασία των δικαστικών λειτουργών. Αυτό εμπόδισε 7 στου 10 δημοτικηγόρου να μπορούν να κάνουν κανονικά τη δουλειά του. Δηλαδή, ούτε ανεξάρτητη νομική αρρωγή οι πολιτικοί κρατούμενοι είναι στο έλεος της κυβέρνησης. Δεν μπορούν να βρουν υπεράσπιση στην εκδίκαση της υπόθεσής τους. Η ανεξάρτητη δικηγορία λοιπόν είναι επίσης κάτι πολύ σημαντικό όταν ε, θέλει ένα διαφωνούντας να υπερασπιστεί τον εαυτό του σε ένα ε, δικαστήριο τη χώρα. Αυτό έχει ξεκινήσει από το 2017 στη χώρα, πρέπει κάτι να κάνουμε. Ευχαριστούμε. Η Επιτροπός, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτέ. Να σας ευχαριστήσω και αυτή τη δυνατότητα να συζητήσουμε και πάλι αυτή την κατάσταση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Αζερμπαϊτζάν. Ακολουθούμε την κατάσταση με μεγάλη προσοχή, όπως και εσείς, και τις τρέχουσες εξελίξεις σε ό,τι αφορά και την υπόθεση του κυρίου Μαχμένα Χουσέινοφ. Αυτό το είχαμε ήδη επισημάνει από το 2017. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω την ευκαιρία αυτή για να σας πω τι έχουμε κάνει ε, για το θέμα αυτό πρόσφατα. Μετά από το διάβημα λοιπόν της ε, αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χάρη στη συνεργασία των ε, αρχών του Αζερβαϊτζάν, η Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία μαζί με πέντε μέλη της αντιπροσωπείας επισκέφθηκε τον κύριο Χούσινεφ στην φυλακή και έτσι καταφέραμε να διαπιστώσουμε ότι η ζωή του δεν είναι σε άμεσο κίνδυνο. Λαμβάνει ιατρική φροντίδα και έχει σταματήσει την απεργία πείνα. Παρ' όλα αυτά, πιστεύουμε, όπω και εσεί, ότι οι κατηγορίε που του απαγγέλθηκαν ε, δεν είναι αξιόπιστε και θα πρέπει να ελεγχθούν. Είμαστε φυσικά ενήμεροι, όπω είπε κάποιο από εσά, ότι λαμβάνουν χώρα και άλλε απεργίε πείνα ακτιβιστών. και παρακολουθούμε τι υποθέσει του μέσω των δικηγόρων, μέσω των υπηρεσιών και ξέρουμε ότι έχουν ε, λάβει επισκέψει και από τον Ερθρό Σταυρό. Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει αρκετό βάρο ε, στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αζερβαϊτζάν και στον πολιτικό μα διάλογο με, τις, ε, με τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων και συναντήσεων υψηλού επίπεδου με εκπροσώπου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των οργανώσεων, του κράτου κτλ. Πέρσι τον Ιούλιο τονίσαμε ότι το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών αποτελούν κλειδί για τις σχέσεις μας. Η νέα Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση και Αζερβαϊτζάν που είναι υπό διαπραγμάτευση θα περιλαμβάνει δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, κράτος δικαίου και καλή διακυβέρνηση καθώς και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών. Είμαστε ε, φυσικά ενήμεροι και αντιλαμβανόμαστε τα βασικά, τις βασικές απειλές ε, κατά των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Αζερμπαϊτζάν και πιστεύουμε ότι μέσω του διαλόγου, μέσω των διαπραγματεύσεων για τη νέα συμφωνία θα πρέπει να έχουμε ανοιχτές διόδους επικοινωνίας για να υπάρχει δυνατότητα αλληλό σεβασμού και αυτό θα ευνοήσει και τις δύο πλευρές του Αζερμπαϊτζάν. Και ενώ συνεχίζουμε τη δέσμευσή μας με τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν, συνεχίζουμε να, να συνεργαζόμαστε και με τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανεξάρτητους δημοσιογράφους, ακτιβιστές και το καθεξής. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να θέτουμε το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ελευθεριών σε όλους μας τους διαλόγους και κυρίως ε, στην επόμενη συνάντηση για τα θέματα δικαιοσύνη ε, και ανθρωπίνων δικαιωμάτων 5 ε, Φεβρουαρίου στον Πακού. Και θα παρακολουθήσουμε και την υπόθεση του κυρίου Χωσέινοβα συγκεκριμένα και των άλλων δημοσιογράφων και της κυρίας Ισμαήλοβα. Και φυσικά θα συνεχίσουμε ε, τον διάλογο και μαζί σας ασφαλώς για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ε, ολοκληρώθηκε η συζήτηση για αυτό το θέμα και όπως γνωρίζετε η ψηφοφορία θα ακολουθήσει σήμερα αργότερα. Ε, και προχωρούμε στο επόμενο θέμα, το οποίο είναι η συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σουδάν. Ε, το λόγο έχει ο κύριος Τάνοκ για 1,5 λεπτό για να αρχίσει η συζήτηση. Πληθωρισμός 122%. Ε, η κυβέρνηση κόβει ε, τα επιδόματα για τα καύσιμα και για τα τρόφιμα. Ο κόσμος έχει εξεγερθεί και αυτό δεν μας ε, εκπλήσει. Ξεκίνησε ενός διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας και ε, ε, των ε, προβλημάτων που δημιουργούνται με τις ουρές για να πάρει ο κόσμος ψωμί. Και τώρα έχει γίνει ένα κίνημα κατά της κυβέρνησης. Η αντιπολίτευση είναι διχασμένη. Ο πρόεδρος Μπασίρ που κυβερνάει 30 χρόνια προσπαθεί να κρατηθεί στην εξουσία που έχει αρπάξει ακυρώνοντας τη διάρκεια της θητείας και καθιστώντας την απεριόριστη απόκριση αυτή ε, που οδήγησε 40 πολίτες ε, άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους και 2 με 3 χιλιάδες άνθρωποι έχουν ε, συλληφθεί και κρατούνται. Θα πρέπει ο κύριος Μπασίρ να εγκαταλείψει την εξουσία και έχει και το ε, φοβερό τίτλο να είναι εν ενεργεία ηγέτης κράτους με δύο εντάλματα σύλληψης του Διεθνούς Δικαστηρίου να εκκρεμούν εις βάρος του. Ε, πολύ ε, διαβόητος. Θα πρέπει λοιπόν να τερματιστεί αυτή η κατάσταση σε αυτή την περιοχή της Αφρικής. Η κυρία Βερζιά για τρία λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλά ψηφίσματα έχουμε ήδη εγκρίνει για το Σουδάν. Το τελευταίο ήταν το Μάρτιο του 2018 για την ε, ε, σύλληψη του ε, Μαχμούτ Αλιώσμα που ε, είχε παλάβει και το βραβείο Ζαχάροφ το 2007. Ε, ε, είναι διαβητικός και ανησυχούν οι συγγενείς του για τη σύλληψη αυτή από τις διαβόητες μυστικές υπηρεσίες. Για άλλη μια φορά δυστυχώς συζητούμε. 2.000 άτομα έχουν συλληφθεί από τις 19 Δεκεμβρίου του 2018. Δεκάδες νεκροί για να μην μιλήσουμε για τα βασινιστήρια. Ε, από το 2013 γίνονται ε, συνεχώς ε, διαδηλώσεις, κυρίως στη Χαρτούμ. Μέχρι τώρα για λόγους οικονομικούς, γιατί έχασαν τους πόρους από το πετρέλαιο όταν διχοτομήθηκε το Σουδάν. Πάνω από 120% είναι ο πληθωρισμός δεύτερος παγκοσμίω και αυξάνονται συνεχώς τα προϊόντα πρώτης ανάγκης σε μια χώρα που έτσι κι έχει προβλήματα από ελλείψεις. Για να μην μιλήσουμε για τον προϋπολογισμό, 70% είναι στρατιωτικές δαπάνες εις βάρος των υπολείπων υγεία και παιδείας κυρίως. Το Δεκέμβρη, αφού τριπλαστιάστηκε η τιμή του ψωμιού, έγιναν οι πρώτες διαδηλώσεις που ε, εκτός της πρωτεύουση και πήγαν σε όλη τη χώρα, εξαπλώθηκε αυτό ε, ως και στον Ταρφούρ όπου ε, ε, ακόμα σοβούν οι Τζιντζαντζάουι και ε, οι γνωστές καταστάσεις. Πολύ γρήγορα τα αιτήματα γίνανε πολιτικά. Ελευθερία, δικαιοσύνη ζητούν και να τερματιστεί το καθεστώς του Μπασίρ ο οποίος έγινε συνηθισμένος στις προκλήσεις και θέλει τώρα να αλλάξει και το Σύνταγμα για να κατέβει ξανά υποψήφιος. Ενώ εδώ και 29 χρόνια είναι πρόεδρος και κρεμούν και πολλά εντάλματα εις βάρος του από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ε, σοβούν οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συλλαμβάνονται ε, οι ε, και από το Δεξιό Κόμμα και από το Κομμουνιστικό Κόμμα που ε, τόλμησαν να δώσουν τα γραφεία τους για να γίνουν διαδηλώσεις, αντιπολίτευσης και συγκεντρώσεις μια εβδομάδα ε, τώρα γίνονται ε, και απο, αποκορύφωμα θα είναι σήμερα μια μεγάλη πορεία στην Χαρτούμ. ζητούμε να αρθούν οι συμφωνίες που έχουμε κάνει με το Σουδάν για τη μεταναστευτική πολιτική καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Μα πώς μπορούμε να συνεργαζόμαστε με αρχές που καταστέλουν τον κόσμο και του ζητούμε να έρχονται και εδώ στα κέντρα κράτησης και να ε, ταυτοποιούν τους πολίτες τους ή τους δίνουμε κάποιο εξοπλισμό που μπορούν να χρησιμοποιούν κατά του λαού και στον Ταρφούρ μάλιστα. Θα πρέπει να αναθεωρήσουμε κάθε χρηματοδότηση για να σταματήσει αυτή η υποκρισία. Τέλος, Θέλω να εκφράσω εξ ονόματο ομάδα μου τη Ενωτική Αριστερά την απόλυτη αλληλεγγύη μου με όλου εκείνου που σήμερα θα διαδηλώνουν στου δρόμου ε, του Σουδάν, ε, διακινδυνεύοντα τη ζωή του. Ευχαριστώ, η κυρία Βαλέρο. Δύο μισή λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχά να μιλήσω για τι αρνητικές αυτέ ε, διαδικασίε. Πιστεύω ότι αυτά θα πρέπει να επιτραπούν. Όταν φυσικά η κυβέρνηση αυξάνει τόσο πολύ τι τιμέ για βασικά τρόφιμα, είναι λογικό να γίνονται τέτοιε διαμαρτυρίε. Και αυτέ οι διαμαρτυρίε ε, έχουν ε, λάβει χώρα από την Ήπετρο στα χωριά μέχρι και την πρωτεύουσα του Χαρτούμα. Είναι λογικό ότι υπάρχει τέτοια διαμαρτυρία κατά του Πρόεδρου Μπασίρη, ο οποίο εδώ και 29 χρόνια είναι στην εξουσία. Θα πρέπει να υπάρξει ένα διάδοχο. Όσοι εργάζονται στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στη χώρα έχουν αναφέρει 45 εκτελέσει ήδη για άτομα τα οποία βγαίνουν και διαμαρτύρονται. Και η μέθοδοι που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση, πώ καταπνίγει τι βίες αυτέ ε, τις ε, διαμαρτυρίες αυτές με βίαιο τρόπο και τους πολιτικούς αντιπάλους. Το Σουδάν λοιπόν και θα πρέπει να ακολουθήσει και το διεθνές δίκαιο. Αυτό δεν συμβαίνει σήμερα. Τα διεθνή αυτά πρότυπα λοιπόν θα πρέπει να ακολουθούνται σε ό,τι αφορά και τις συλλήψεις, τις καταδίκες. Επίσης, σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση ατόμων, τα βασανιστήρια που διαβάλλουν χώρα στις φυλακές, δεν μπορούμε να τα δεχτούμε αυτά σε καμία χώρα. Και επίσης, τίθεται και το θέμα του ημερολογίου για την εξαγωγή εκλογών. Το 2020 υποτίθεται ότι το συνταγματικό, το συνταγμα δεν επιτρέπει να ξανακατεύει σε εκλογέ ο πρόεδρο. Παρ' όλα αυτά, όμω προσπαθεί, όπω σε πολλέ άλλε χώρε φυσικά γίνεται αυτό, να κατέβει, να αλλάξει το σύνταγμα. Και χρησιμοποιεί του νομικού που πρόσχονται σε αυτό να Ζητείτε λοιπόν η ε, υπηρεσιακή κυβέρνηση και νέα προκήρυξη εκλογών σε νέα ημερομηνία. Έχω λίγο χρόνο και να κάνω και μία ακόμα ερώτηση για το ψήφισμα αυτό, το ψήφισμα το οποίο βασίζεται σε τρέχοντα περιστατικά παράδεκτα. Όταν ε, μιλάμε για την κατάσταση του Σουδάν, για μένα ως πράσινη, είναι πραγματικά λυπηρό το γεγονός ότι διαπιστώνω ότι τα μέσα τα οποία ήδη έχουν ληφθεί εδώ και δεκαετίες έχουν ε, αρνητικές επιπτώσεις και στο περιβάλλον. Είναι πραγματικά φρικτές οι καταστάσεις από τις οποίες ο κόσμος προσπαθεί να ξεφύγει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα το λόγο έχει ο κ. Πάετ για Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Παρά τις ε, εβδομάδες διαμαρτυριών στο Σουδάν και τις κλήσεις για παρέτηση του πρόεδρου Αραμάν Πασίρε έχει προταθεί για νέες εκλογές ε, και για νέα θητεία ο πρόεδρος Μπασίρα ε, για το 2020. Το PCP, το κυβερνόν κόμμα, δήλωσε ότι η ηγεσία του κόμματος θα αλλάξει μόνο στις εκλογές. Αυτό φυσικά δεν το έχουμε δει ακόμα. Και το γεγονός είναι ότι ο Μπασίρη είναι ο μοναδικός ε, αρχηγός κράτους που διώκεται, κράτος που διώκεται από το Διεθνές Δικαστήριο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, γενοκτονία, εθνοκάθαρση στον Ταρφούρ και παρόλα αυτά παραμένει ελεύθερος, συνεχίζει τα εγκλήματά του. Τον καλωσορίζουν δε και τόσα πολλά κράτη. Με ανοιχτά αγκαλίε. Ινδία, Κίνα, Κατάρα, Σαουδική Αραβία και πολλέ ακόμα εξακολουθούν να επιτρέπουν στον Μπασίρ να έρχεται στη χώρα τους, τον καλωσορίζουν αντί να τον συλλάβουν. Και λόγω της αδράνειάς τους ε, μπορεί το καθεστώς Μπασίρ να συνεχίσει την ατιμορρυσία του και να επιτίθεται σε πολίτες. Και γι' αυτό λοιπόν ε, βλέπουμε τις τελευταίες αυτές δράσεις του Μπασίρ, όπου 37 τουλάχιστον άτομα έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 800 συνελήφθησαν αυτό το κύμα βίας και καταπίεσης από τις αρχές. Μαζικές εκτελέσεις, συλλήψεις κατά των ακτιβιστών, ε, δημοσιογράφων, ε, δασκάλων, δικηγόρων. Ο Μπασίρ λοιπόν θα πρέπει να κριθεί για τα εγκλήματα που του καταλογίζονται. Και στις τελευταίες από τις διαμαρτυρίες θα πρέπει λοιπόν να προσαχθεί στη δικαιοσύνη. Έχει έρθει η ώρα το Σουδάν να επικεντρωθεί στην ε, στον τερματισμό τη καταπίεση και τη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να αναλάβει το ρόλο τη ω μια υπεύθυνη κοινωνία. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρο. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Κιέγγια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στο επίκεντρο της προσοχής μας έχει έρθει τώρα το Σουδάν, μια από τις πιο εκτεταμένες αφρικανικές χώρες. Οι πρόσφατες ειδήσει από το Σουδάν έχουν αποδειχθεί πολύ δυσάρεστες. Ενώ μεγάλο μέρο του κόσμου ε, γιόρταζε την πρωτοχρονιά, οι κάτοικοι του Σιδάν βγήκαν στους δρόμους και τις πλατείες της χώρας, ε, διαμαρτυρώμενοι για την μείωση της αγοραστικής τους δύναμης. Λόγος της διαμαρτυρίας ήταν οι αυξήσεις στις τιμές πρώτα της βενζίνης, μετά του ψωμιού, του οποίου με προεδρικό διάταγμα τριπλασιάστηκε η τιμή. Στη χώρα ξεκίνησαν οι διαμαρτυρίες και οι διαδηλώσεις, αλλά έτσι τίθεται να αμφιβόλω η πολύ λεπτή ισορροπία με τα, της κοινωνίας γιατί είναι επισφαλή ο καθημερινό βίο των πολιτών. Η οικονομική συγκυρία δεν είναι ευνοϊκή για τη χώρα. Παρόλο που έχει πολλού πόρου, το Σουδάν προχωρά στην ιστορία με, μεταξύ περιόδων σχετική ηρεμία και άλλων που είναι ιδιαίτερα δύσκολε για του πολίτε. Ε, περνούν λοιμού ε, λόγω τη κακοδιαχείριση τη κυβέρνηση και πολλέ φορέ υπάρχουν κοινωνικέ συγκρούσει με ε, αντίδραση των δυνάμεων δίωξη τη χώρα την καταστολή. Το τίμημα το πληρώνουν όχι μόνο όσοι διαφωνούν με την κυβέρνηση του Σουδάν, αλλά και οι διαμαρτυρώμενοι ίδιοι. Το Σουδάν επιβεβαιώνει την θλιβερή πραγματικότητα της καταστολής των πολιτικών ελευθεριών. Ε, δεν επιτρέπει τους απελπισμένους πολίτες να εκφραστούν. Η κυβέρνηση του Χαρτούμ θα πρέπει να θυμηθεί ότι έχει ευθύνε για την ανάπτυξη της ίδιας της χώρας. Μόνο με την καλλιέργεια των οικονομικών δραστηριοτήτων της χώρας και τη δημιουργία ενός υγιούς πολιτικού κλίματος μπορεί να καταπραϊνθούν αυτές οι κινήσεις διαμαρτυρίας. Είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε και το ρόλο του πολιτικού διαλόγου που θα πρέπει να ε, διοργανωθεί ιδίω μετά τον συνασπισμό των κομμάτων αντιπολίτευσης. Πρέπει να αποφυλακιστεί και ο νικητής του βραβείου Ζαχαρόφ, Σαλή Μαχμούντοσμάν και όλοι όσοι θέλουν να συλλογίζονται και να σκέφτονται ελεύθερα. Ε, καθηγητές του Πανεπιστημίου του Χαρτούμ, δημοσιογράφοι και προσπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για να υπάρξει ένα πιο δημοκρατικό Σουδάν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κέλλαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το Σουδάν είναι ανεξάρτητο εδώ και 63 χρόνια. Περίπου πριν από 30 χρόνια ο Αλμπασίρ ανέλαβε την εξουσία. Ε, απαγόρευσε τη δημιουργία πολιτικών κομμάτων και προέβλεψε το μουσουλμανικό νόμο ως βασικό νόμο της χώρας από το Σύνταγμά της. Έχει μείνει πρόεδρος από το 1993. Το Σουδάν λοιπόν έχει γίνει μονοκομματικό ε, κράτος ε, και αργότερα στη δεκαετία του 1990 αναφέρθηκε και καταγράφηκε ως ένα κράτος που χρηματοδοτούσε τρομοκρατικές οργανώσεις. Από την ίδια την κυβέρνηση. Ε, εδώ και κάποια χρόνια ο ε, Μπασίρ προσχέθηκε να διοργανώσει εκλογές. Το ακούμε από το εδώ και χρόνια μάλλον, το 2018 ε, εμποδίστηκε η διοργάνωση ελεύθερων εκλογών ως προς την ελευθερία του τύπου. Είναι το Σουδάν 174ο στη λίστα των χωρών και τι επιδόσει του στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, πριν τι γιορτέ ξεκίνησαν διαμαρτυρίε για τι αυξήσει τη τιμέ τη βενζίνη και του ψωμιού. Όμω, όσοι διαμαρτύρονται κατά το πολιταρχικού καθεστώτο και καλούν ε, τον ε, πρόεδρο Αλμπασίρ να παρατηθεί, ε, έχουν υποστεί διώξει. Όπω είπα, κατά την εξουσία εδώ και 30 χρόνια. Είναι εκατοντάδε οι άνθρωποι που έχουν συλληφθεί λόγω των διαμαρτυριών του και έχουν φυλακιστεί και πασανιστεί. Ο νικητή του γραφείου Ζουχάρεφ Σαλή συνελήφθη πάλι πριν από 9 μέρε. Είναι γνωστό, άγνωστο μάλλον που βρίσκεται. Ε, το Σουδάν είναι η τέταρτη χειρότερη χώρα ως προς την στάση της ε, έναντι των χριστιανών. Καταδικάζουμε λοιπόν την, τη δίωξη των χριστιανών από τις κρατικές αρχές, το κλείσιμο των εκκλησιών, τους υποχρεωτικούς προσελητισμούς των χριστιανών στη μουσουλμανική θρησκεία. Ε, ένα άλλο γεγονό που θα πρέπει να έχουμε υπόψη και το οποίο αναφέρθηκε πριν από λίγα λεπτά είναι ότι ο Αλ Μπασίρ είναι ο μόνο ασκών καθήκοντα αρχικού κράτου που ε, έχει, ε, θα έπρεπε να προσέλθει στο Διεθνέ Δικαστήριο για εγκλήματα κατά τη ε, ανθρωπότητας και γενοκτονίας στην περιοχή του Νταρφούρ. Θα πρέπει ε, να πάψει να κυβερνά αυτός ο διεθνής παρείας στη χώρα ε, και έτσι να γίνεται αντιληπτική χώρα του. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, λάβει υπόψη αυτέ τι σοβαρέ διαμαρτυρίε που έχουν γίνει στη χώρα και να ζητήσει την άμεση απελευθέρωση του κυρίου Οσμάν και όλων των ακτιβιστών και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει όλοι οι πολίτε να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και να υπάρξει πραγματική ελευθεροτυπία στη χώρα. Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την είπατε πρόσωπο να ε, καταδικάσουν δημοσίω και με αυστηρότητα την κατάσταση στο Σουδάν, απαιτώντα από την κυβέρνηση να μεταβάλει τη στάση τη, να πάψουν οι μαζικέ συλλήψει Επίσης, καλούμε για μια ε, επικαιροποίηση του συστήματος εξαγωγών και ε, του συστήματος ασφάλειας που χρησιμοποιείται για τις εμπορικές μας σχέσεις με το Σουδάν. Επίσης, να φροντίσουμε και η τεχνολογία παρακολούθησης του διαδικτύου να λειτουργεί σωστά στη χώρα. Θα χρειαστεί υποστήριξη για τους ακτιβιτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του εκπροσώπους τη κοινωνία των πολιτών στο Σουδάν μέσω από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Κύριε συνάδελφε, και τώρα... Ε, ε, ήσασταν εσείς ο τελευταίος συντάκτης του ψηφίσματος. Ακολουθούν οι πολιτικές ομάδες. Ο κύριος Δεχόφσκι, για δύο μισή λεπτά, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το Σουδάν θα μπορούσε να είναι μια πολύ ωραία χώρα, εάν στη χώρα αυτή ε, δεν υπήρχε ε, αυτό το ολοκληρωτικό καθεστώς. Δεν είναι η μόνη χώρα, αλλά δεν είναι και η πρώτη φορά που συζητούμε την περίπτωση του Σουδάν. Πολύ συχνά ε, υπάρχουν πάρα πολλές αδικίες. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω όλες τις περιπτώσεις που ακούσαμε, γιατί θα ήταν πολύ μακρά η συζήτηση. Η ανεξιθρησκεία και οι θρησκευτικέ ελευθερίες αποτελούν ουτοπία στη χώρα αυτή. Είναι χιλιάδες ε, οι μαρτυρίες που έχουμε και οι αποδείξεις για βασανισμούς, οι βασανιστήρια. Μόλις πρόσφατα συζητούσαμε ε, για τον Πέτερ Γιάσκο, ένα Τσέχο εργαζόμενο ε, στην ανθρωπιστική βοήθεια που είχε φυλακιστεί για ένα χρόνο. Και μας εξηγούσε τι γίνεται με τους μη μουσουλμάνους ή με τους άθεους. Ε, τι βασανιστήρια υφίστανται, αυτές τους εικονικούς πνιγμούς, το waterboarding και άλλα σκανδαλώδη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αντιδράσει και να ασκήσει πίεση ε, στο Σουδάν να σταματήσει αυτές τις πρακτικές. Είναι πολλοί υποστηρικτές μας και χάρη σε αυτούς ε, καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια κατάσταση όπου να αλλάζει σιγά σιγά η ατμόσφαιρα και το κλίμα που επικρατεί ε, στον πληθυσμό. Αυτό ισχύει για άλλε χώρε. Για το Σουδάν ακόμα δεν έχει γίνει πραγματικότητα. Θα πρέπει να στείλει και είπατε εκπρόσωπο ένα πολύ σαφέ μήνυμα προ το Σουδάν ότι δεν πρόκειται να ανεχθούμε τι αδικίε και ε, τα δεινά που υφίσταται ο λαό. Οι καθημερινοί άνθρωποι. Δεν μπορούμε εμείς να συνομιλούμε με προέδρους που δολοφονούν τους ίδιους τους πολίτες της χώρας τους και παραβιάζουν ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν πρόκειται ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει τέτοιες καταστάσεις ή τέτοιους ανθρώπους, πολιτικούς ηγέτες υποτίθεται που επενδύουν τα χρήματά τους σε άλλες χώρες, όχι στη δική τους. Και αυτά θα πρέπει να τα γνωρίζουν και άλλες χώρες. Ότι το Σουδάν είναι το χειρότερο δικτατορικό καθεστώς που υπάρχει στην Αφρική και όποιος το υποστηρίζει δεν είναι εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Και τώρα το λόγο έχει από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες ο κύριος Κριστέα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα πρέπει να πω ότι οι πρόσφατες διαδηλώσεις ήταν ειρηνικές από το Δεκέμβριο σε όλο το Σουδάν. Δεν είναι μόνο στη Χαρτούμ, σε όλη τη χώρα δικαίως διαμαρτύρονται οι πολίτες για τις αυξήσεις των τιμών στα καύσιμα και στα τρόφιμα και για τις ελλείψεις. Ε, αυτές οι διαδηλώσεις κατεστάλησαν με τρόπο πάρα πολύ βίαιο από τις δυνάμεις ασφαλείας. Η ελευθερία της έκφρασης κανονικά είναι ε, συστατικό της δημοκρατίας. Θα πρέπει η κυβέρνηση ε, του Σουδάν να αντιμετωπίσει αυτά τα δίκαια αιτήματα του λαού και να μην καταφεύγει στη βία για να λύνει το πρόβλημα βία η οποία οδήγησε σε θάνατο 40 ατόμων, μεταξύ αυτών και παιδιά, με αυθαίρετες συλλήψεις αγνώστου αριθμού διαδηλωτών, ε, μεταξύ αυτών και φοιτητών, ε, σπουδαστών, ε, δημοσιογράφων. Θα πρέπει να φεθούν ελεύθεροι όλοι οι κρατούμενοι και να γίνουν ανεξάρτητες έρευνες. Και όσοι αποδειχθούν ένοχοι να προσαχθούν στα δικαστήρια. θα πρέπει και οι μυστικές υπηρεσίες, μάλλον οι δυνάμεις ασφαλείας της χώρας, να ελέγχονται για τη συμπεριφορά τους. Να ε, επιτρέπονται επισκέψεις ε, των μελών των οικογενειών των δικηγόρων ε, στους κρατουμένους. Τα βασανιστήρια και οι πρακτικές αυτές είναι απαράδεκτες. Καλούμε την κυβέρνηση να τερματίσει κάθε είδους βίαιη συμπεριφορά και να προχωρήσουν ε, αν υπάρχει εγγύηση για δίκαιες δίκες μόνο οι διώξεις αυτές. Ο κύριος Δεμές Μάκερ. Ε, Συνάδελφοι, την προηγούμενη εβδομάδα ο Economist δημοσίευσε τον ετήσιο δίκτυο για τη δημοκρατία και το Σουδάν ως αυταρχικό καθεστώς είναι κάτω-κάτω σε παγκόσμιο επίπεδο. Το η χώρα αυτή δεν μοιάζει καθόλου στη δημοκρατία. Δεν υπάρχει ουσιαστικά εύρυθμα ε, ε, λειτουργών κράτου και αρχέ. Ε, οι πολιτικέ ελευθερίε είναι ουσιαστικά ανύπαρκτε. Η διεθνή κοινότητα έγραψε πολλέ πολλέ εκθέσει για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα, ωστόσο δεν αλλάζουν τίποτα. Αυτό που λειτουργεί είναι τα στρατεύματα ασφαλεία και η εθνοφρουρά που με βίαιο τρόπο καταπνίγουν τι διαμαρτυρίε του κόσμου στου δρόμου του 14ου Μπασίρα σε ό,τι αφορά την οικονομική ανασφάλεια ασφάλεια που υπάρχει και ε, χάρη στο, λόγω του καθεστώτος του χαρτούμα. Στις ε, πρόσφατες λοιπόν ε, διαδηλώσεις ήταν δεκάδες οι νεκροί και εκατοντάδες οι τραυματισμένοι. Είναι γνωστές αυτές οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί το καθεστώς κατά των ακτιβιστών δημοσιογράφων και μελών της αντιπολίτευσης. Ουσιαστικά όμω ο κόσμο λέει ή «Λοιπόν, που θα πεθάνουμε και θα πεθάνουμε από την πείνα στα σπίτια μα, θα βγούμε στου δρόμου. Αυτό ακούγεται στου δρόμου. Θα πρέπει λοιπόν το Κοινοβούλιο να επιλέξει την πλευρά που θα υποστηρίξει και να εκφράσει την υποστηρίξη του για τους του, του, την κοινωνία των πολιτών και για το λαό, ο οποίο διαρκώ κοινοποιείται κινητοποιείται στο Σουδάν κατά των παραβιάσεων αυτών των ανθρώπινων δικαιωμάτων γιατί δεν μπορεί να υπάρξει καλύτερη κοινωνία με τον κύριο Μπασίρ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα θα πάρει το λόγο ο κύριο Καστάλντο. Ευχαριστώ. Ο λαός θέλει να φύγει η κυβέρνηση. Θα πρέπει να σταματήσουν να γεμίζουν οι φυλακές του Χαρτούμ με τη χρήση ε, δακρυγόνων, μολότοφ ε, και άλλων μέσων δίωξη και καταστολής των πολιτών. Οι πολίτε τη χώρα ζητούν την παρέτηση του Προέδρου και την αλλαγή τη κυβέρνηση. Χάο επικρατεί στη χώρα. Όχι μόνο γιατί οι αστυνομικέ δυνάμει, αλλά γιατί και παραστρατιωτικέ και μυστικέ υπηρεσίε βιαίω επιτίθονται στου πολίτε και του διαμαρτυρόμενου. Ο απολογισμό είναι τραγικό. 45 νεκροί. Ε, και εκατοντάδε ε, που φυλακίστηκαν την περασμένη μόλι εβδομάδα. Ε, και όλα αυτά για την αλλαγή ένα καθεστώτο, αυτού του Αλμπασίρ, που κυβερνάει εδώ και 30 χρόνια θα πρέπει ε, οι καταγγελίες, μάλλον οι κατηγορίες του για γενοκτονία και εγκλήματα κατά ανθρωπότητα στον Ταρφούρ να οδηγήσουν στην πλήρη ε, αναστολή της ε, προεδρικής του θητείας και τη διοργάνωση εκλογών στη χώρα πολύ σύντομα. Το 2020 ο κ. Οσμάν, νικητής του βραβείου Ζαχάροφ και οι 20 φοιτητές ε, του Πανεπιστημίου του Νταρφούρ συνελήφθησαν τον Δεκέμβριο ξανά. Θα πρέπει να ζητήσουμε κάθε ε, πάυση τη μορφή συνεργασία εμπορική, πολιτική, οικονομική με τη χώρα αυτή για να πάυσει αυτή η σφαγή, άδικη σφαγή των πολιτών τη χώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος, η κυρία Αρνωτή, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. ο Βάτιγκερ, ο Αρή Λεβί μάλλον, ε, σε ένα δελτίο που κυκλοφόρησε ε, που κυκλοφόρησε το πέρσι ε, κατηγορούσε την ε, χώρα για την ε, κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από το Δεκέμβριο εκατοντάδες συνελήφθησαν ε, από τις αρχές του Δεκεμβρίου και θυμίζει αυτό την εξέγερση των κίτρων γυλαίκων στη Γαλλία κατά του Πρόεδρου Μακρόν. Είναι δεκάδες τα θύματα στο Σουδάν και στη Γαλλία όμως είναι εκατοντάδες. Και επίσης η παρέτηση του Υπουργού ήταν στη Γαλλία, Καστανέρη ήταν μία αρχή. Θα πρέπει ε, στην Ευρώπη να δούμε ότι οι Ισλαμιστές συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος. Γι' αυτό λοιπόν συνάδελφοι κάποιε φορές εκπλήσω με τα κηρύγματα που κάνουμε στους άλλους. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ασχοληθεί με το τι γίνεται κάτω από τη μύτη του αντί να ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα σε άλλες υπήρους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Χέτσμαν, για να είμαι Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κυρίε και κύριοι. Οι διαμαρτυρίε οι οποίε λαμβάνουν χώρα στην ε, τελευταίο μήνα γίνονται όλο πιο αιματηρέ και όλο και πιο βίαιες. Η μεγάλη πλειονότητα των Σουδανέζων ζουν σε συνθήκες απόλυτης ένδυα. Έχουν λιγότερο από ένα δολάριο την ημέρα για να επιβιώσουν. Δεν είναι λοιπόν περίεργο το γεγονό ότι οι τιμέ των τροφίμων που αυξήθηκαν οδήγησαν του Σουδανέζους στου δρόμου. Και οι προτινόμενε αλλαγέ στο Σύνταγμα προκειμένου ο πρόεδρο Μπασίρ να ανακριχθεί πρόεδρο διαβίου ο ίδιο πρόεδρο, ο οποίο έχει κατηγορηθεί για βίαιε παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για γενοκτονία. Είναι λοιπόν καθήκον τη Ευρωπαϊκή Ένωση να καλέσει τι αρχέ του Σουδάν να σταματήσουν τη χρήση βία και να απελευθερώσουν τους φυλακισμένους ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να σταματήσουν τη δίωξη των χριστιανών και άλλων θρησκευτικών ομάδων. Η ελευθερία έκφρασης περιορίζεται, η πρόσβαση στο διαδίκτυο περιορίζεται επίσης σε ό,τι αφορά και την απαγόρευση που πρέπει να υπάρξει στι εξαγωγέ προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη βασανιστήρια. Ευχαριστώ και το λέω έχει η κυρία Κουόρτ για δύο λεπτά. Την προηγούμενη εβδομάδα ο Μαρ Ελχάζε, Σουδανό δημοσιογράφος που μένει στη Λίβερπουλ, στη δική μου περιφέρεια, ε, ήρθε σε επαφή μαζί μου γιατί ανησυχούσε για την κατάσταση στη χώρα της. Μου λέει λοιπόν η κυρία αυτή ότι ο κόσμος ε, είναι αντιμέτωπος με ανεφρεγμένων επίπεδα βίας σε ό,τι αφορά τις διαμαρτυρίες κατά της ε, καταπίεσης του Μπασίρη. Πυροβολισμοί στον αέρα. Έχει λοιπόν ατράνταχτα αποδεκτικά στοιχεία για την κατάσταση αυτή. Η κατάσταση λοιπόν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του blogger κυρίου Άλλη, ο οποίο πυροβολήθηκε από σνάιπερ το Δεκέμβριο και πέρασε 10 μέρε στην εντατική. Δύο ημέρε μετά απήχθη από το ίδιο του το σπίτι, από τι ιδανικέ Αρχέ Ασφαλεία και πλέον κρατείται ε, σε απάνθρωπες συνθήκες χωρίς δυνατότητα Είμαι πολύ ανήσυχη για την κατάστασή του. Καλό λοιπόν τι αρχέ τη Σουδάν να τον απελευθερώσουν άμεσα, να του δώσουν την ιατρική φροντίδα που χρειάζεται στο εξωτερικό. Επίση, θα πρέπει οι αρχές να ενημερώσουν την οικογένειά του και τον δικηγόρο του για τον, τρόπο, για τον τόπο που κρατείται και να επιτρέψουν επικοινωνία με αυτόν. Η κατάσταση του είναι πολύ ανησυχητική και η κατάσταση των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πολύ ανησυχητικά. Καλούμε λοιπόν την Επιτροπή να επιμείνει προκειμένου να απελευθερωθεί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κόσμο στον Λίβερπουλ που στέκεται στο πλευρό των Σουδανών αυτές τις δύσκολες στιγμές. Δεν θα παραδοθούμε ποτέ σε αυτό το εχθρικό περιβάλλον της Τερίζα Μέη σε ό,τι αφορά τους πρόσφυγες, τους αιτούντες άσυλο και τους μετανάστες. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Κέλλη για 1,5 λεπτό. Uh, Ευχαριστώ. Και πάλι συζητούμε την νυχτρή κατάσταση στο Σουδάν σε σχέση με τις εμελιώδεις ελευθερίες. Ο κόσμος άρχισε να διαμαρτύρεται για την ακρίβεια και κατέδυσε να διαμαρτύρεται κατά της κυβέρνησης δεν υπάρχει ελευθερία ε, του συνέρχεστε, αυθαίρετες ε, ε, συλλήψεις απέναντι σε ειρηνικούς διαδηλωτές. Επίσης καταδικάζω απερίφραστα την κράτηση του Σαλή Μοχάμετ Οσμάν, ο οποίος μάλιστα κρατείται και σε άγνωστο σημείο και καλό να αφαιθεί αμέσως ελεύθερος. Και άλλοι ακτιβιστές αντιμετωπίζουν αντίστοιχες παραβιάσεις και θα πρέπει και αυτοί να αφαιθούν ελεύθεροι. Θα πρέπει επίση να σταματήσουν οι διωγμοί των χριστιανών. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό για το ΕΛΚ, την ομάδα μας που είναι χριστιανοδημοκρατική ομάδα. Ένας ελεύθερος τύπος, ανεξάρτητος, με παλόμενη συζήτηση είναι πυλώνας μιας δημοκρατικής κοινωνία. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ελευθερία. Ε, του τύπου και της έκφρασης και να το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους εξωτερικούς εταίρους της και το Σουδάν για να αφαιθούν οι πολίτες να ε, λειτουργούν στην κοινωνία των ε, πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα και των γυναικών κυρίως παραβιάζονται. Θα πρέπει να καλέσουμε τις αρχές του Σουδάν να σεβαστούν τις διεθνείς υποχρεώσεις τις οποίες έχουν αναλάβει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα κύριος Χάν για δύο λεπτά παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε. Οι πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στο Σουδάν μας ανησυχούν βαθύτατα. Θα πρέπει να απαντήσουμε με κυρώσεις μέχρι να σταματήσει η καταστολή άρχισε ως μια διαμαρτυρία για τις τιμές του ψωμιού και των καυσίμων και πλέον έχει ε, στραφεί κατά του καθεστώτος του Αλμπασίρ που κυβερνάει 29 χρόνια. Οι δυνάμεις ασφαλείας πάταξαν αμήλικτα αυτές ε, τις ε, διαδηλώσεις με πραγματικά πυρά, με δακρυγόνα κλπ εκατοντάδες ε, ε, πολιτικοί ηγέτες, δημοσιογράφοι, απλοί πολίτες ε, διώκονται και κινδυνεύει να γίνει ακόμα πιο αιμοσταγής η κατάσταση γιατί προσπαθεί να γαντζωθεί στην εξουσία με κάθε τίμημα ο Αλμπασίρ. Το δικαίωμα του συνέρχεστε, του συνεχερίζεστε και τη έκφρασης θα πρέπει να γίνεται σεβαστό, Όπω ορίζει το διεθνέ Δίκαιο, να απελευθερωθούν αμέσω όλοι οι κρατούμενοι και να διερευνηθούν όλες οι καταγγελίες για αυθαίρετες συλλήψεις και κρατήσεις και οι να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι εκκρεμεί ακόμα και ένα ένταλμα σύλληψη του, κατά του κυρίου ε, Μπασίρ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και για γενοκτονία. Χαίρομαι με αυτά που λέτε. Ε, πρόεδρε ε, και Επιτροπέ, αλλά δεν αρκούν η διεθνή κοινότητα θα πρέπει να σταματήσει να εθελοτυφλεί στα όσα κάνει για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων το Σουδάν. Και τέλος κύριε Πρόεδρε, έχει έρθει η ώρα να επιβάλλουμε ε, κυρώσει απέναντι στους υπευθύνου για τις σοβαρέ παραβιάσεις και να αναθεωρήσουμε τη διμερή μας συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ. για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε, Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Παρά τα γεγονότα ότι έχουν γίνει κάποιες αλλαγές στην νομοθετική διαδικασία, τα πρόσφατα γεγονότα που περιέλαβαν τη μασική χρήση βίας, η κατάσταση στο Σουδάν εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ επισφαλής, γιατί συνεχίζει να αρνείται βασικά και θεμελιώδη δικαιώματα και συμφωνώ ότι θα πρέπει τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη να παίξουν μεγαλύτερο ρόλο στην περιοχή και να ερευνήσουν αυτέ τι περιπτώσει καταπίεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίση, θα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να υπάρξει μεγαλύτερη πρόσβαση των δεύτερων οργανώσεων για την παροχή ανθρωπιστική βοήθεια σε αυτού που τη χρειάζονται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίση θα πρέπει να κάνει πιο πολλές προσπάθειες σε ό,τι αφορά την ελευθερία έκφρασης μέσω των εξωτερικών μέσων και εργαλείων που έχει στη διάθεσή της και να ενισχύσει τους ακτιβιστές και όσους προσπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη και το ενδεχόμενο να μειώσουμε τους πόρους προς το Σουδάν αν χρειαστεί σε περίπτωση που οι πόροι αυτοί χρησιμοποιούνται με τέτοιο τρόπο. Απαράδεκτο. Τέλος. Πλήρης διαφάνεια θα πρέπει να υπάρχει σε ό,τι αφορά τα έργα ασφάλειας σε συνεργασία με το Σουδάν και όλες ε, οι δραστηριότητε που προγραμματίζονται με ευρωπαϊκούς πόρους. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Περνάμε τώρα στη διαδικασία Catch the Eye. Ο κύριος Φαρία είναι ο πρώτος ε, που θα λάβει το λόγο. Παρακαλώ, έχετε ένα λεπτό κύριε Φαρία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Όταν ε, ξεκίνησαν οι μαζικές ε, διαμαρτυρίες πριν από ένα μήνα, λόγω της αύξηση τεράστια των τιμών ε, Προκάλεσε δυστυχών, ε, δυστυχώς η καταστολή και δίωξη των διαδηλωτών που ήταν κατά της διαφθοράς. Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση συνεχίζει να εφαρμόζει αυθαίρετες συλλήψεις και διώξεις και μάλιστα είχαμε ακόμη και θανάτους και πολλαπλές κατάφορε παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά ακτιβιστών και απλών πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μείνει προσιλωμένη στι βασικέ τη αξίε. και να συνεχίσει να ασκεί πιέσει προς τον πρόεδρο Μάραλ Μπασίρ και στους υπόλοιπου ε, υπευθύνου παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να σταματήσει την καταστολή και να ε, απελευθερώσει ακτιβιστές μεταξύ των άλλων και τον ε, Μαχμούτ Αλίος Μάνα, τον δικηγόρο και προβραβείο Ζαχάροφ 2007. Επίσης θα πρέπει να σταματήσει την καταστολή Αλμπασίρ και θα μπορούσαμε να ασκήσουμε πίεση διακόπτοντας οποιαδήποτε χρηματοοικονομική βοήθεια προς την κυβέρνηση Αλμπασίρ. Ο κύριος Ρόπες Αγγιλάρ, ένα λεπτό κι εσείς. Κύριε Επίτροπε, κύριε Επίτροπε, στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία είχα την ευκαιρία και την ε, χαρά να λάβω μέρος σε μία αποστολή παρατήρηση εκλογών στο Σουδάν και εκεί πραγματικά είδα η σώμαση τη τεράστια λαχτάρα του Σουδανικού λαού για δημοκρατία. Ε, και δυστυχώς επανειλημμένως έχουμε ε, συζητήσει κατάφορες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σουδάν υπό την πίεση του Πρόεδρου Αλμπασίρ, που διώκεται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και προωθεί παρόλα αυτά μια συνταγματική αναθεώρηση που θα οδηγήσει σε περαιτέρω παράνομες κρατήσεις των ακτιβιστών που πραγματικά κόπτονται και διαφέρονται για το κράτος δικαίου στο Σουδάν και τη δημοκρατία. Είπατε ότι εκπρόσωπος Μογκερίνη ε, έκανε κάποια διαβίβατα, αλλά εσείς που είστε υπεύθυνοι για το εμπόριο, αρμόδιο επίτροπος για το εμπόριο, να Μεριμνήσεται ώστε να επιβληθούν κυρώσει σε αυτή την απολύτω απαράδεκτη συμπεριφορά του καθεστώτο Αλμπασίρ. Μια συμπεριφορά που απάδει ριζικά από τι ε, αξίε και αρχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε και εμεί. Ο κύριο Μαριά έχει το λόγο. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η καταπίεση είναι στην ημερήσια διάταξη στο Σουδάν με την περίφημη Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και Ασφαλείας να συλλαμβάνει, να ασκεί βία, να βασανίζονται οι ακτιβιστές οι σπουδαστές και όσοι τολμούν να διαδηλώσουν. Ε, όλα αυτά έχουν ενταθεί βεβαίως μετά την οικονομική κρίση η οποία υπάρχει παρότι το σουδάν είναι μια πλούσια χώρα στην πράξη ο λαός αγωνίζεται για ένα κομμάτι ψωμί. και φυσικά ο πρόεδρος ο αλ μπασίρ ο οποίος ε, θα πρέπει κανονικά να παραπεμφθεί στο διεθνές ποινικό δικαστήριο προσπαθεί να επεκτείνει τη θητεία του γιατί μόνο έτσι νομίζει ότι θα γλιτώσει από την διεθνή ποινική δικαιοσύνη απαιτείται λοιπόν να ληφθούν μέτρα να επιβληθούν κυρώσεις να καταλάβει ο μπασίρ και η παρέα του ότι δεν μπορεί να εφαρμόζει τον ισλαμικό νόμο δεν μπορεί να εκδιώκει τους αντιφρονούντες δεν μπορεί να εκδιώκει τους χριστιανικούς πληθυσμούς και πρέπει κυρία μάλμστρομ να έχουμε άμεσα μέτρα κυρώσεις κατά του καθεστώτος του σουδάν. ευχαριστώ. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με το σχέδιο ψηφίσματος που θα ψηφιστεί σήμερα. Βλέπω ότι την κατάσταση στο Σουδάν όπως και οι συνάδελφοί μου. Να προσέξουμε κάτι θλιβερό, ότι ξανά μιλάμε για την κατάσταση στο Σουδάν. Ξανά μιλάμε για την καταστολή των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε αυτήν την Αφρικανική χώρα και επιδεινώνεται καθημερινά η κατάσταση. Δεν ξέρω αν υπάρχει λύση. Θα ήθελα να σα ρωτήσω, κυρία Μάλστρομ, τι λέτε, πρέπει να ε, σα ζητήσω να αυξήσουμε τι κυρώσει ε, κατά του καθεστώτο, να μειωθούν οι ενισχύσει κατά του καθεστώτο του Μπασίρ, να κατασχεθούν οι λογαριασμοί τραπεζικοί των μελών του καθεστώτο. Ε, μόνο οι κυρώσει μπορούν να ασκήσουν πιέσει σε αυτό το τρελό καθεστώ αλλά φοβούμε ότι αυτό δεν αποτελεί την πλήρη λύση. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα ψηφίσματα έχουν μεγάλη συμβολική αξία και ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη συμβολική αξία τη μεταφράσει συγκεκριμένα βήματα και μέτρα τα οποία θα ανατρέψουν το καθεστώ του Μπασίρ. Σα ευχαριστώ. Και τελευταίο ο στα πλαίσια του ΚΑΤΣΤΙΑ, ο κύριο Ιτουργάη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα πρέπει να κάνουμε μια ανάλυση της κατάστασης ε, της αφρικανικής αυτής χώρας του Σουδάν. Ανισότητα, έλλειψη πόρων, βιαιότητα, βιοπραγίες, ε, έλλειψη ελευθεροτυπίας, καταστολή του, των πολιτών. Πρόκειται για μια διάγνωση που ισχύει και για άλλες χώρες της Αφρικής, αλλά στο Σουδάν ε, το πολιτικό και κοινωνικό τοπίο είναι όλο και πιο ανησυχητικό. Γιατί η αντιπολίτευση υφίσταται διώξεις και φοβερή καταστολή. Και στις διαδηλώσεις, για τη διάλυση των διαδηλώσεων χρησιμοποιούνται καταστολή βίας. Έχουμε πάνω από 50 νεκρούς, για να μην μιλήσω για τραυματίες. Είχαμε πάρα πολλές ε, ε, βίες ε, εκδηλώσεις στο Σουδάν και θα συνεχιστεί η καταπίεση της αντιπολίτευσης αν δεν αντιδράσουμε. Και πραγματικά είναι μακάβριο το καθεστώ του Αλμπασίρ και συνεχίζει την καταπίεση. Για να μην μιλήσουμε για τι διώξει των χριστιανών ή ε, των ε, άλλων πιστών, άλλων θρησκειών που δεν μπορούν ελεύθερα να ασκήσουν την θρησκευτική του πίστη. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε μέτρα να επιβάλλουμε κυρώσει στο, στον Αλμπασίρ για την άδικη μεταχείριση του λαού που επιβάλλει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Και για να ολοκληρώσουμε θα παρακαλέσω την Επίτροπο κυρία Μάλμστρομ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι. Αξιότιμη Ευρωβουλευτέ. Η κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σουδάν εξακολουθεί να μας ανησυχεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προβληματιζόμαστε κυρίως λόγω της ε, καταπολέμησης ελευθεροτυπίας, της ελευθερίας του συνέρχεστε, του συνεταιρίζεστε, αλλά και της συρρήκνωσης του ζωτικού χώρου της κοινωνίας των πολιτών. Γινόμαστε μάρτυρες αυτής της κατάφορης παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τις τελευταίες εβδομάδες μετά την βία επάντηση της κυβέρνησης του Σουδάν για τις εκτεταμένες διαδηλώσει και διαμαρτυρίες από το Σεπτέμβριο λόγω της αύξησης του κόστου των βασικών αγαθών και της έλλειψης βασικών αγαθών. Η κυβέρνηση απάντησε με σφαίρες από καουτσούκ, με βία καταστολή, με συλλήψεις ακτιβιστών και πάνω από 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και πάνω από 800 εξακολουθούν να είναι κρατούμενοι και είναι ε, κατασχέσει πολλών ε, ε, πρακτοριών ειδήσεων και υπάρχει μεγάλη καταστολή και φραγή των ειδήσεων ώστε να μην ενημερώνονται οι διαδολωτέ. Επίση, χρησιμοποιήθηκαν δακρυγόνα ακόμη και κατά νοσηλευτικού προσωπικού. Και μάλιστα κάναμε δηλώσει και διαβήματα ζητώντα από τη Σουδανική κυβέρνηση να απελευθερώσει δημοσιογράφου, ακτιβιστέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικηγόρου και όλου όσου έχουν ε, φυλακιστεί αυθαίρετα. Επίση, περιμένουμε διεξοδικέ ε, διαλευκάνσει ε, των καταχρήσεων και των θανάτων που έχουν σημειωθεί. Θα πρέπει οι δράστε να δώσουν λόγο για τα έργα του. Επίση, θα πρέπει το καθεστώ να αποφύγει τη χρήση βία ε, για να αποκλιμακωθεί η κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε από την κυβέρνηση του Σουδάν να επιτρέψει το Σουδανικό λαό να ασκήσει το συνταγματικό του δικαίωμα και να εκφέρει ελεύθερα τη γνώμη του χωρί να φοβάται την καταστολή. Επίση, ζητούμε από την κυβέρνηση να εφαρμόσει τις απαραίτητες πολιτικές ε, ε, μεταρρυθμίσεις για να αντιμετωπίσει τα δεινά του λαού και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα. Ε, θα συνεχίσουμε να είμαστε ε, υπέρμαχοι ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών στο Σουδάν και θα στηρίζουμε το έργο τη κοινωνία των πολιτών και των ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων με του διάφορου τρόπου που έχουμε στη διάθεσή μα. Όπω ξέρετε, οι σχέσει μα με το Σουδάν έχουν επηρεαστεί από τη, τα εντάλματα συλλήψη ε, του Διεθνού Ποινικού Δικαστηρίου κατά του Πρόεδρου Αλμπασίρ και ε, την άρνηση του Σουδάν ε, να κρίνει την αναθεωρημένη συμφωνία του Κοτονού. Άρα το Σουδάν δεν είναι πια επιλέξιμο για τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια η χώρα βρίσκεται σε δεινή οικονομική και ανθρωπιστική κατάσταση. Εκτεταμένες συγκρούσεις, αβεβαιότητα στα σύνορα, όλα αυτά επηρεάζουν αρνητικά την κατάσταση στην περιοχή. Και γι' αυτό προβλέψαμε ένα ειδικό μηχανισμό για το Σουδάν με ένα εκατομμύριο ευρώ κονδύλιο πριν από δύο χρόνια για να ε, ευνοήσουμε τον πληθυσμό. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγκρίνουμε την πολιτική ηγεσία και τα μέτρα της, αλλά ε, έχουμε δρομολογήσει αυτό το κονδύλιο μέσω του Trust Fund για την Αφρική, του Καταπιστευματικού Ταμείου Καταπήγου Ανάγκη για την Αφρική, προκειμένου να βοηθήσουμε του πλέον απόρου και ευάλωτου του Σουδάν. Συνεχίζουμε να επισημαίνουμε τις ανησυχίες μας σε όλα τα επίπεδα των επαφών με τις Σουδανικές Αρχές και συνεχίζουμε την ε, υποστήριξή μας προς το μέσο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας και χρησιμοποιούμε τα διάφορα κονδύλια για να προωθήσουμε την ελευθεροτυπία και την διαπαιδαγώγηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Σουδάν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Έχω λάβει έξι σχέδια ψηφίσματος για το θέμα αυτό. Ολοκληρώνουμε τη συζήτηση και διακόπτουμε τώρα μέχρι την ψηφοφορία που θα λάβει χώρα εντός ολίγου. Θα έχουμε ένα σύντομο διάλειμμα μέχρι την έναρξη της ψηφοφορίας. Σας ευχαριστούμε και πάλι για τη συμμετοχή στη συζήτηση και ευχαριστούμε και την Επιτροπό. Good afternoon, colleagues. The voting... Καλησπέρα, συνάδελφοι. 12 Ήταν ε, στο πρόγραμμα να ξεκινήσουμε στις 12. Τώρα έχουν περάσει οι 12 ακριβώ και σας δίνω ένα-δύο λεπτά μόνο για να καθίσετε στις θέσεις σας και να ξεκινήσουμε. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και τους ε, συναδέλφους που με βοηθούν στο να εξασφαλιστεί η ησυχία και η ηρεμία στην αίθουσα. Έχουμε αρκετές ψηφοφορίες μπροστά μας. Πριν, δώσω, πριν προχωρήσω στις ψηφοφορίες, δίνω το λόγο στην κυρία Πύρη που με παρακάλεσε να μιλήσει πριν από την άνοιξη των ψηφοφοριών. Παρακαλώ κυρία Πύρη. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι. Ο Ολλανδός δημοσιογράφος σήμερα απρόβλεπτα απελάθη από την Τουρκία και διερωτώ με αν για άλλη μία φορά έχουμε να κάνουμε με ένα παράδειγμα για, του τρόπου με τον οποίο η Τουρκία αντιμετωπίζει τους δημοσιογράφους και παρακαλώ τον Πρόεδρο Ταγιάννη να έρθει σε επαφή με τις τουρκικές αρχικές και να ζητήσει γιατί η δημοσιογράφος αυτή έχει απέλαθει. Γιατί εξηγήσει πέραν ε, κάποιε ασαφεί περί δεσμών με τρομοκρατική οργάνωση δεν έχουν δοθεί και πάλι για άλλη μια φορά τίθενται ζητήματα σε σχέση με την αντιμετώπιση του τύπου και την ελευθεροτυπία στην Τουρκία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ βεβαίως και σας στηρίζει ολόκληρο το Κοινοβούλιο. Ως πρώην δημοσιογράφος και εγώ στηρίζω το αίτημά σας. Κύριε Γουλφ, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Μια και είμαστε στα διαδικαστικά. Καλό θα ήταν να λέμε σε ποιο άρθρο του κανονισμού αναφερόμαστε για να μην καθυστερούν και οι διαδικασίες. Αυτό πολλές φορές μας το έχουν πει και εγώ έχω αντίστοιχες παρεμβάσεις να κάνω όπως ε, της ε, κυρίας που μίλησε μόλις τώρα. Μπορείτε να μας ανημερώσετε λοιπόν επικαλούμενοι ποιο άρθρο ε, έλαβε το λόγο η συνάδελφος για να μπορώ και εγώ να το επικαλούμε στο μέλλον και να ομιλώ. Η Πρόεδρος, βεβαίως θα παρακαλέσω τις υπηρεσίες να έρθουν σε επαφή μαζί σας κύριε Γουλφ. Ο κύριος Νόσνιτς, ο συνάδελφος και γείτονά σας ζητεί το λόγο, παρακαλώ. Ε, ε, Την Τρίτη, η κυρία Μπιλμπάο Μπαραντίκα μίλησε απρεπώς είπε ότι έξι ομιλητές ε, για την επέτειο του ευρώ ήταν άντρες. Ε, τουλάχιστον ε, στη, στην όψη, αλλά μπορεί να νιώθουν ε, και τη γυναική τους φύση. Δεν θα πρέπει να κάνει τόσο φαλοκρατικά σχόλια για τέτοια άνηση μεταχείριση. Πρέπει να είναι ελεύθεροι άνθρωποι να νιώθουν όπως θέλουν and their first report relates to Azerbaijan, notably the case of Έχουμε να ψηφίσουμε λοιπόν τώρα με το πρώτο θέμα που αφορά το Αζερβαϊτζάν. Κυρία Χάρμς, έχετε το λόγο. Έγινε πολύ καλή διαπραγματεύση για το ψήφισμα αυτό με τους αδέλφους. Όλοι μαζί υπογράψαμε το ψήφισμα. Πρέπει ωστόσο να σας υποβάλω δύο προφορικές τροπολογίες, τεχνικού χαρακτήρα μόνο, για να είναι απολύτως σωστό το ψήφισμα. Και θα ήθελα να ζητήσω το λόγο για τα σημεία B και C του ψηφίσματος, αλλά αν συμφωνείτε μπορώ τώρα να σας εξηγήσω τις δύο ε, τεχνικές αυτές προφορικές τροπολογίες και σας παρακαλώ να κάνετε δεκτές τις εξής αλλαγές. Στο σημείο B του ψηφίσματος, ο Μουχμάν Χοζέινοφ που αναμένεται να αποφυλακιστεί το Μάρτιο του 2019 είναι αντιμέτωπος με μια πρόσθετη ποινή φυλάκισης 5 έως 7 ετών ε, που του επιβάλλεται όχι δυνάμει το άρθρο 352, αλλά δυνάμει το 372. Αυτή είναι η πρότασή μας και παρακαλώ να την υποστηρίξετε. Και επίσης η δεύτερη, η οποία αφορά την, την επίσκεψη της ε, αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης στη φυλακή όπου κρατείται ο Χουσέινοφ, επίσκεψη η οποία έλαβε χώρα όχι στις 10 Ιανουαρίου, αλλά στις 11 Ιανουαρίου. Ύστερα από τα όσα δεν είπε ο Επίτροπος ε, στην ε, συζήτηση, ε, δηλαδή ότι ο Χουσεϊνόφ μετά την επίσκεψη αυτή της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης διέκοψε την απεργία πείνας ο Χουσεϊνόφ, η απεργία απεργία ήταν κομμάτι του ψηφίσματο. την επικαλούμαστε στο ψήφισμα, θέλω να ε, καταστήσω σοφέ, σαφές ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί η διακοπή αυτή τη απεργία πείνα από την οικογένεια και του δικηγόρου του Χουσέινοφ. Αυτά ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη στι δύο αυτέ τεχνικέ αλλαγέ. Ευχαριστώ λέει η, Πρόεδρε, Οι Πρόεδρος. Υπάρχουν ε, αντιρρήσει ω προ τι δύο αυτέ προσαρμογέ του κειμένου. Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται και σας ευχαριστώ κοινό ψήφισμα έξι πολιτικών ομάδων για το Σουδάν. Υπέρ. Κατά. Αποχές και εγκρίνεται. πρόγραμμα συνδρομής για την ε, πυρηνική για τον παροπλισμό του πυρηνικού σταθμού υπέρ κατά πέρας προφορίας μάλλον εγκρίνεται έκθεση πυρήνσκη ετήσια έκθεση για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ονομαστικά Πέρας. Εγκρίνεται έκθεση Σβόποντα, διασυνοριακέ αιτήσει επιστροφών έργων τέχνη και πολιτιστικών αγαθών που λελετήθηκαν σε περίοδο ενόπλων συγκρούσεων και πολέμων. Ονομαστικά, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση Ρέγνερ Απόφαση τη Επιτροπή Νομικών Θεμάτων για την άνοιξη διαπραγματεύσεων επί τη βάση τη εκθέσεω τη κυρία Ρέγνερ για τι διασυνοριακέ μετατροπέ συγχωνεύσει και διασπάσει. Θέλει καλή να λάβει το λόγο. Πολύ καλά. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται λοιπόν η απόφαση της Επιτροπής. Μπορείτε να ξεκινήσετε τις πραγματεύσεις αμέσως στο επόμενο θέμα. Ψηφοφορία για την απόφαση της Επιτροπής Αλίας για την άνοιξη διαπραγματεύσεων επί τη βάση της εκθέσεως κύριε Ρακαρσία, δέσπιση πολιτικού σχεδίου για τις ελευθερικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης αυτοπελαγικών αποθεμάτων στη Δυτική Μεσόγειο. Θέλει κανεί το λόγο. Παρακαλώ η συνάδελφος, κυρία Κιλέρα. Ευχαριστώ ηρεμία. Θα σας αρέσουν αυτά που θα πω. Έχουμε την ευκαιρία, ψηφίζοντα ναι στην εντολή, να έχουμε για πρώτη φορά ένα σχέδιο αληφ... διαχείριση διαχείρισης για τη Δυτική Μεσόγειο. Γι' αυτό ζήτησα την εντολή. Κάναμε τεράστια προσπάθεια ε, με τις συμβαστικές τροπολογίες. 24 ε, εγκρίναμε μέχρι την τελευταία στιγμή και μάλιστα ανα, αναβάλαμε την ψηφοφορία στην Επιτροπή για να συγκεντρώσουμε μεγαλύτερη συνένεση. Τα καταφέραμε και με την ψηφοφορία αυτή θα έχουμε την ευκαιρία για πρώτη φορά να έχουμε ένα σχέδιο ελευτική διαχείρισης για τη Δυτική Μεσόγειο, ένα σφαιρικό πλαίσιο διαχείρισης της Ελίας. Γιατί αν πούμε όχι στην εντολή, δεν θα έχουμε ε, σχέδιο διαχείρισης για την Ελία στη Μεσόγειο. Ψηφίστε ναι λοιπόν. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Όχι, ψηφίζουμε λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία ονομαστικά. Πέρας. Εγκρίνεται. Και μπορούμε να ξεκινήσουμε σε Μπορεί να ξεκινήσει η Επιτροπή Διαπραγματεύσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Και η επόμενη έκθεση. Βλέπω ότι είστε καλοδιάθετοι σήμερα. Μακάρι, όλη τη μέρα. Κυρία Γκάρτια Σαπάρ, Ρουμπιάλ και Σαρβάμα ήταν η επόμενη έκθεση. Προστασία του προπολογισμού τη Ένωση στην περίπτωση γενικευμένων λήψεων όσον αφορά το κράτο δικαίου στα κράτη-μέλη. Κύριε Σαρβάμα, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ένα από τα πιο σημαντικά και κρίσιμα στοιχεία που απαιτούνται για την ε, διαφύλαξη της ε, δημοκρατίας σε κάθε κράτος, σε κάθε κράτος μέλος είναι το κράτος δικαίου. Η υπονόμευση του κράτους δικαίου είναι πάντα επικίνδυνη γιατί ανοίγει το δρόμο για την αποδυνάμωση άλλων στοιχείων ενός δημοκρατικού κράτους και γι' αυτό ψηφίζουμε την έκθεσή μας. Επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω πως ο κανονισμός αυτός βρίσκεται τη νομική του βάση στον δημοσιονομικό κανονισμό, το άρθρο 322 και όχι το άρθρο 7 της συνθήκης. Στόχο έχει δηλαδή την προστασία του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού από γενικευμένες ελλείψεις ε, όσον αφορά το κράτος δικαίου. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό για την έκθεση και την πρότασή μας που πρέπει να αντιληφθείτε είναι ότι πρέπει να υπάρξει και θα υπάρξει το ίδιο σύνολο δημοσιονομικών συνεπειών για οποιοδήποτε κράτος μέλος θα έθετε σε κίνδυνο το κράτος δικαίου ή θα υπονόμευε το κράτος δικαίου. Ευχαριστώ κύριε Σάρβαμα. Ψηφίζουμε λοιπόν ε, την ε, πρόταση για απόρριψη της πρότασης Επιτροπής. Πέρας. Απερίφθη. Κύριε Σάρβαμα, έχετε προφορική τροπολογία να προτείνετε. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η προφορική τροπολογία έχει ως εξής η πρόληψη και τιμώρηση φοροαποφυγής και η εξασφάλιση σωστών ε, συνθήκων ε, λειτουργίας ε, της διοίκησης με τη διαγραφή των όρων και φορολογικού ανταγωνισμού. Αυτή είναι η πρότασή μας. Ο φορολογικός ανταγωνισμός είναι αρμοδιότητα των πρώτων μελών και γι' αυτό δεν έχει θέση μέσα στην έκθεσή μας. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν αντιρρήσεις? Μάλιστα. Υπάρχουν. Μπορείτε να ξανακαθίσετε αγαπητοί συνάδελφοι. Και σας διαβάζω ακριβώς το κείμενο για να μην μπερδευτούμε. Έχουμε να κάνουμε τις τροπολογίες της αρμόδιας επιτροπής 128, 133, 37 με 44, 45 με 68 και τη 41 όπως αρχικά έχει κατατεθεί υπέρ κατά επαληθεύω Πέρας. Εγκρίνεται τροπολογία 36 ονομαστικά παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται 72 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη 29 υπέρ. Κατά. Αποχ... Εγκρίνεται. 81 υπέρ. Θέλετε να επαληθεύσω την 29. 81 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη 73 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη 69 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη 45 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 62 υπέρ όχι 82 διορθώνει η πρόεδρος, 82 υπέρ κατά. Αποχές απερίφθη 70 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη 71 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη 57-61 αντί υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 76, 77 καταπίπτουν, 79 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 80 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Πρόταση της Επιτροπής συνολικά, ονομαστικά πάντα. Πέρας. Και εγκρίθηκε. Κυρία Καρδιά Σαμπάλ Ρουμπιάλ για να σχολιάσει παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ για την βρή ε, αυτή υποστήριξη. Θα ζητήσω λοιπόν το Κοινοβούλιο να αναπέμψει την υπόθεση στην Επιτροπή την Αρμόδια για τις Δημοσιονομικές Διαπραγματεύσεις με βάση το άρθρο 59α, ε, δεδομένου ότι έχουμε αυτές τις εκκρεμότητες. Ευχαριστώ πολύ. Ψηφίζουμε αυτό λοιπόν υπέρ κατά. Αποχές και εγκρίνεται, αναπέμπεται στην καθήλυνα αρμόδια για τις διαπραγματεύσεις επιτροπή και έκθεση Giggold τώρα θέσπιση του προγράμματος φυσικάλης για τη συνεργασία στον τομέα της φορολογίας τροπολογία παριθμών 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 και 3 ονομαστικά άρχεται okay. πέρας εγκρίνεται Η 1CP2 καταπίπτει και τώρα ψηφίζουμε την πρόταση της Επιτροπής. Πέρας. Εγκρίνεται. Παρακαλώ τον κύριο Κίκολτ να λέω το λόγο. Δεν ζήτησα το λόγο, Πρόεδρε, αλλά πρέπει προφανώς να αναπευθεί στις δύο οργανικές διαπραγματεύσεις. Βεβαίως και αυτή την πρόταση την ψηφίζουμε παρακαλώ υπέρ, κατά αποχές και γίνεται δεκτή κύριε Γκίγκολτ και η πρόταση αυτή και προχωρώ στην επόμενη έκθεση. Έκθεση Βαλέρο. Θέσπιση του προγράμματος Δικαιώματα και Αξίες. 113-114 μαζί ονομαστικά. Πέρασε. απερίφθησαν οι άλλες, η ομάδα ακόμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκαν 21 ονομαστικά υπέρ, άρχεται ψηφοφορία μάλλον συγγνώμη, πέρας. Εγκρίνεται 73. Πρώτο τμήμα ονομαστικά. Πέρας. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα ονομαστικά. Πέρας. Και απερίφθη. Πρόταση της Επιτροπής ονομαστικά. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται κυρία Βαλέρο. Κυρία Βαλέρο, ζητώ συγγνώμη λέει πρόεδρος. Έχετε το λόγο. Θα ήθελα να αναπευθεί στην Επιτροπή το θέμα για διοργανικές διαπραγματεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 59.4. Αυτά. Σας ευχαριστώ κυρία Βαλέρο. Ψηφίζουμε το ΡΕΠΕΡ. Κατά αποχές εγκρίνεται και το θέμα αναπέμπεται ξανά προς διαπραγματεύσεις. Προχωράμε στο επόμενο θέμα, επόμενη έκθεση. Ούρτιτσεφ, Ευρωπαϊκό Μηχανισμό στον τομέα τη ποινική ασφάλεια, συμπληρώνει το μηχανισμό γειτονία ανάπτυξη διεθνού συνεργασία. Τροπολογία 1.47 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνονται. Τροπολογία 48 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Πρόταση τη Επιτροπή. Ονομαστική ψηφορία. Άρχεται. Πέρα. Εγκρίνεται. Πηγαίνουμε τώρα στην έκθεση τη κυρία Κόμισον αφού καταπολέμηση καθυστερήσεων πληρωμών σε εμπορικέ συναλλαγέ, παράγραφο 4. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ. Έλεγχο για το δεύτερο τμήμα, παρακαλώ. Πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Ονομαστική κλίση. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Συγγνώμη, ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Το ψήφισμα με ονομαστική κλίση που άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στην έκθεση κυρία Κάπελ, ετήσια έκθεση για τι χρηματοδοτικέ δραστηριότητε Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το ψήφισμα, αν κλίση» που υπάρχετε. Πέρα. Εγκρίνεται. Επόμενη έκθεση για, για διαφοροποιημένη ολοκλήρωση, έκθεση Ντιράν, ονομαστική κλίση, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται συνάδελφοι, σας ευχαριστώ. Τελική έκθεση του κυρίου Λάινερ και της κυρίας Τόμ, παράγραφος 8, πρώτο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 16, πρώτο τμήμα, ονομαστική κλίση, άρχεται. Πέρας. εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ονομαστική κλίση άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Το ψήφισμα ονομαστική κλίση άρχεται. Πέρας. Και εγκρίνεται συνάδελφοι και σας ευχαριστώ. Παρακαλώ συνάδελφοι να αποχωρήσετε για να προχωρήσουμε στις επεξηγήσεις ψήφου. Μπορούμε να συνεχίσουμε μέχρι στις 14 και 45. Πάμε στην έκθεση Μπέγκε. Η κυρία Κέρτον Ντάρλινγκ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Δεν βλέπω την κυρία Κέρτινγκ Ντάρλινγκ στην αίθουσα. Ο κύριος Σόσνιεφ, έχετε το λόγο. Νομίζω ότι τηλεφωνάει τώρα. Ο κύριος Ζάχαντριλ, για ένα λεπτό, για επεξήγηση ψήφου για την έκθεση Μπέγκε. Δεν καταφέρνω να μας κάνουν σε επεξηγήσεις ψήφου. Πάμε σε άλλη έκθεση και επιστρέφουμε σε αυτήν. Ναι. Συνάδελφος Χάουαρτ, επεξήγηση ψήφου για την έκθεση Φερνάντες Γκουτιγέρο για το πρόγραμμα Invest EU. Έχετε το λόγο. Uh, um, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Όταν συναντώ κάποιου που συμμετέχουν στα προγράμματα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεως λένε ότι χρειάζεται απλούστευση. Έχουμε κάποια απλούστευση σαν αποτέλεσμα τη εκθέσεως. Έχουμε μείωση όσον αφορά τα ακρονίμια πρέπει να χρησιμοποιούμε. Έχουμε νέο καθεστώ ε, διαχείριση και έχουμε 13 υπηρεσίε που συναθρίζονται σε ένα σημείο επαφή. και αυτή η απλούστευση επίση δίνει κάποια ευελιξία ευελιξία για να μπορούμε να βρούμε το κατάλληλο πρόγραμμα. 38 δισεκατομμύρια λίρες και οι αγγίσεις και άλλα 9,5 δις από εθνικούς και περιφερειακούς εταίρους είναι αρχή. Και τελικά το αποτέλεσμα είναι η επένδυση που είναι 650 δις. Αυτή είναι η εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι μια επένδυση που δίνει χρήματα ε, που δεν μπορεί να δώσουν οι άμεσες εμπορικές επενδύσεις. Ο ιδιωτικό και εμπορικός τομέας μαζί επενδύουν στο Invest Euro και αυτό αφορά την βοηθά στη μελλοντική ανάπτυξη. Ευχαριστώ κυρία Μακοβέη. Ευχαριστώ. Τώρα, αυτή τη στιγμή, το, τα επίπεδα προστασία των επενδύσεων δεν ανταποκρίνονται στις διευθυντικές ανάγκες τη ευρωπαϊκή Ενώσεως. Και οι αλλαγέ δεν είναι μακροπρόθεσμες τεχνολογική φύσεω. Δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στις κοινωνικές αλλαγέ και τις γενικότερες αλλαγέ που χρειάζονται συνεχή στήριξη. Γι' αυτό στηρίζω το Ταμείο Invest EU, διότι θα βοηθήσει να αναπτυχθεί η έρευνα, και να αναπτυχθεί και η ψηφιοποίηση, που αυτό θα οδηγήσει σε απασχόληση, θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και θα πετύχουμε και τους στόχους της Συμφωνία των Παρισίων για την αλλαγή του κλίματος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να επενδύσουμε στον πολιτισμό, στην τεχνολογία, στην παιδεία, την επαγγελματική κατάρτιση. Ένα σημαντικό δικαιούχο. Ε, αυτού του προγράμματο είναι και θα πρέπει να είναι η Ρουμανία, διότι έχει πολύ μεγάλου ανθρώπινου πόρου. Αυτού του τομεί η Ρουμανία. Ευχαριστώ στην έκθεση ΜΑΤΟ για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Συγγνώμη, για να σα ακούσω πρέπει να ενεργοποιήσετε το μικρόφωνο σα. Είχα ζητήσει επεξήγηση ψήφου και για την έκθεση για την Κεντρική Αμερική και για τη συγκεκριμένη έκθεση ΜΑΤΟ. Δεν σα βλέπω όμω τον κατάλογο για την Κεντρική Αμερική και το άφησα για αργότερα για να επανέλθουμε γιατί έδωσα το λόγο σε τρει συναδέλφου και κανένα δεν ανταποκρίθηκε. Ναι, αλλά εγώ ήμουν εδώ. Ναι, αλλά δεν σα είδα στον κατάλογο. Θα περάσουμε στην επόμενη έκθεση και θα επανέλθουμε. Ε, πριν που σα έδωσα το λόγο κύριε Σωσνιές, μιλούσατε στο τηλέφωνο. Μια στιγμούλα θα επανέλθουμε αργότερα, σε ένα λεπτό. Γιατί πρέπει να περάσουμε στην επόμενη έκθεση που είναι έκθεση ΜΑΤΟ για την ετήσια έκθεση Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο κύριος Μορέλ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εορτάσαμε την 20η ε, ε, επέτειο της ε, ύπαρξης του ευρώ και καλό θα ήταν να κάνουμε μια κριτική και στην ετήσια έκθεση της, του 2017 για την ΕΚΤ. Σίγουρα η ποσοτική χαλάρωση συνέβαλε αποφασιστικά στη διαφύλαξη της ακεραιότητας της Ευρωζώνης και ε, να προστατεύσει τις χώρες του Νότου που υπέστησαν τα πάδινα. Οι πολιτικές όμως που ασκηθήκαν ε, ήταν ανεπαρκείς. Ε, και αντί να ζητήσουμε επεκτατικές πολιτικές, επενδυτικές, για να επιτύχουμε μεγαλύτερη σύγκληση στην Ευρωζώνη, η πρόταση της έκθεσης επανέρχεται στο κλασικό δόγμα το διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που είναι απαραίτητες, που ξέρουμε παρόλα αυτά ότι ε, ρημάζουν ε, περιφέρειες και χώρες όπως έγινε. Αν είχαν προταθεί ε, κάποιες λύσεις για τις αποκλήσεις στην Ευρωζώνη με επενδύσεις, με τις μεταφορές και, πέραν, και αγοράς κρατικών ομολόγων από την ΕΚ, δυστυχώς τίποτα δεν έγινε. Πιστεύω ότι η Ευρώπη αξίζει μια πολύ καλύτερη αντιμετώπιση. Ευχαριστώ. Επανέρχομαι τώρα στην πρώτη μας έκθεση για την Κεντρική Αμερική θα δώσω το λόγο στην κυρία Κέρτορ Ντάρλινγκ, αλλά δεν τη βλέπω στην Ολομέλεια. Οπότε περνάμε στο δεύτερο ομιλητή, τον κύριο Σόσνιε, που έχει το λόγο για ένα λεπτό για την αιτιολόγηση ψήφου για την έκθεση για την Κεντρική Αμερική. Θα σα ε- εξηγήσω γιατί καταψήφισα την έκθεση Μπόγκε. Πρόκειται για έκθεση που αφορά την εμπορική συμφωνία με την Κεντρική Αμερική. Αναφέρεται ε, το θέμα της ισότητας φύλων στα θέματα της εμπορικής συμφωνίας. Δεν νομίζω ότι ε, έχει αυτό νόημα, γιατί αναφέρεται και τα θέματα του διαχωρισμού των δύο φύλων. Ε, διαχωρισμός των φύλων. Τότε να πούμε ότι το εμπόριο είναι γυναίκα. Έχει γυναικείο φίλο, όπως ο Κοπέρνικος, ο Γαλιλαίος όλοι αυτοί ήταν γυναίκες, αν θέλετε. Να το δούμε έτσι. Ο κύριος Ζαχαραντήλα Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ε, δεν θα μπορούσα ούτε και εγώ να υπερψηφίσω την έκθεση. Παρόλο που συμφωνώ με την αξιολόγηση παρόμοιων εμπορικών συμφωνιών, αλλά πέρασε δυστυχώ μια τροπολογία που δεν με βρίσκει σύμφωνο. Την ιδέα τη επιβολή κυρώσεων κατά τη διαδικασία αξιολόγηση. Δεν θεωρώ ότι η κυρώσει είναι αποτελεσματικό τρόπο για τη βελτίωση τη εφαρμογή μια εμπορική συμφωνία. Φυσικά θα πρέπει να ανησυχούμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στι χώρε αυτέ ή για την προστασία του περιβάλλοντο. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι λύση οι κυρώσει. Υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί και μέσα για να εξασφαλίσουμε την εφαρμογή. Και πρόεδρο τη Επιτροπή Εμπορίου. Ήμουν ανέκαθεν κατά των κυρώσεων και αυτό δεν μπόρεσα να υπερψηφίσω την έκθεση Βέγκε. Ο κύριο Χάναν. Ευχαριστώ κυρία Αντιπρόεδρε. Κλείνει το μικρόφωνο δυστυχώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια προσέγγιση για για την Κεντρική Αμερική που δείχνει μια οργάνωση που ενδιαφέρεται για την εξαγωγή της ιδεολογίας της, ε, όπως κάθε επαναστατικό καθεστώς, στην Αυστρία, στη Ρωσία, Μπολσεβίκη για παράδειγμα, ε, και καλεί τις υπόλοιπες ε, περιοχές του κόσμου να την αντιγράψουν όλες οι συμφωνίες με την Κεντρική Αμερική στηρίχθηκαν στην αρχή ότι θα πρέπει να υπάρχει περιφερειακή ολοκλήρωση παντού. Δηλαδή να γίνεται διαπραγμάτευση μεταξύ διαφόρων μπλοκ. Και δεν θέλουν εμπορικές συμφωνίες με μεμονά κράτη. Και η Κεντρική Αμερική εξωθήθηκε στο να δημιουργήσει υπερεθνικές συμφωνίε, όπω το Παρλασέν, που είναι ένα υπερεθνικό κοινοβούλιο, και καταλαβαίνω γιατί γίνονται όλα αυτά. Φαντάζομαι μερικοί πιστεύουν ότι η περιφερειακή σύνδεση και ολοκλήρωση είναι ο καλύτερο τρόπο για να προωθεί ο κόσμο προ αυτή την κατεύθυνση. Κι όμω ε, η δυσάρεστη αλήθεια είναι ότι το αντίθετο συμβαίνει. Το 1950 όταν συστήθηκε η ΕΟΚ ήταν πολύ λιγότερε χώρε. Τώρα είμαστε πολύ περισσότερε. Ένα λεπτό προβλέπεται για τι επεξηγήσει ψήφου. Δεν θα δεχτώ υπέρβαση χρόνου. Έκθεση Τόρβαλτ. Ο κύριο Μορέλ, νομίζω, έχει, έκθεση, έχει επεξήγηση ψήφου στην έκθεση Τόρβαλτς για την Τραπεζική Ένωση. Για την Τραπεζική Ένωση, συμφωνούμε. Ναι, ωραία. Μπορώ να ξεκινήσω την αιτιολόγηση ψήφου. Δέκα χρόνια μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση που ρήμαξε την παγκόσμια οικονομία, η Τραπεζική Ένωση εξακολουθεί να είναι ημιτελής. Οι συστημικές τράπεζες δεν διαλύθηκαν και εξακολουθούν να απειλούν τις κοινωνίες μας λόγω της χρόνιας αστάθειάς τους. Και γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση νέας κρίσης οι χώρες θα υποχρεωθούν να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να κοινωνικοποιήσουν τις απώλειες του χρηματοπιστωτικού συστήματος όπως έγινε το 2008. Οπότε οι υποσχέσεις για τη λύση ε, της κρίσης του 2008 δυστυχώς αθετήθηκαν και έχουμε τη μειωστή έκθεση για την κατάσταση της Τραπεζικής Ένωσης που δεν μας καθησυχάζει καθόλου και μάλιστα ουσιαστικά είναι απόδειξη της αποτυχίας ε, της δεκαετούς εφαρμογής της νεοφιλελεύθερης οικονομίας. Θέλουμε μια ουσιαστική λύση στο πρόβλημα. Θα πρέπει να διαχωρίσουμε τα μιευτήρια από τις επενδυτικές τράπεζες και θα πρέπει να διακόψουμε αυτή την ε, δημοσιονομική λιτότητα. Θα πρέπει να ρυθμίσουμε περαιτέρω και τη σκιώδη τραπεζική που έχει αποσταθεροποιήσει την παγκόσμια οικονομία. Δυστυχώ δεν έχουμε σταθεί στο ύψο των περιστάσεων και αν δεν τα καταφέρουμε θα βρούμε μπροστά μα μια νέα κρίση. Ευχαριστώ. Επόμενη συμφωνία για την εφαρμογή της Εμπορικής Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Κολοβίας και Πέρου, αλλά η κυρία Κέρτον Ντάρλινγκ απουσιάζει. Περνάμε στην κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017. Η κυρία Σόιντροβα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Έχουμε μία κατάσταση για το πρόγραμμα Value και την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο, κύριε Αντιπρόεδρε. Θα ήθελα να σας εξηγήσω γιατί δεν μπόρεσα να υπερψηφίσω την έκθεση Τερή Όλοι ενδιαφερόμαστε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και παρόλο που οι ευρωπαϊκές χώρες είναι δημοκρατικές και έχουν στηρίζουν τις βασικές αρχές, δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε στις δάφνες μας. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα. Δυστυχώς η έκθεση υπερβαίνει αυτό το πλαίσιο. Δεν συμφωνώ με τη σύσταση που ζητά κύρωση της συνθήκης της Κωνσταντινούπολης, γιατί αυτό είναι απόφαση εθνικής κυριαρχίας για τα κράτη-μέλη. Απορρίπτω λοιπόν τη βασική ιδέα της έκθεσης ότι οι υπηρεσίες που αφορούν ε, τα την αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα ε, συμπεριλαμβανομένης και της νομικής άμβλωσης είναι από τα, ε, τα έγκληματα της βάρος των γυναικών. Ευχαριστώ. Εγώ, σοσιαλιστής και ε, το αποκορύφωμα του 2018 ήταν η θέσπιση του Ευρωπαϊκού Πυλώνα ε, Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Είναι από τις θεμελιώδεις αξίες και αρχές μας. Και είναι από τα πρώτα πράγματα που σκέφτονται οι ξένοι όταν μιλούν για την, πολιτική, την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώ, βέβαια δεν είναι τέλεια τα πράγματα ούτε και εντό του οίκου μα. Και το πιο ανησυχητικό σε αυτή την έκθεση είναι τα θεμελιώδη δικαιώματα ε, των μειονοτήτων και οι διακρίσεις που υφίστανται. Δυστυχώ, εξακολουθούν να ισχύουν σε πολλέ χώρε. Η ρητορική του μίσου, ε, δυστυχώ, θέτει σε κίνδυνο πολλού Ευρωπαίου πολίτε και ανεπαρκείς πολιτικές ε, ενσωμάτωσης κοινωνικής ένταξης ε, να αποβαίνουν βάρος των μεταναστών. Ελπίζω λοιπόν να διαβρύνουμε την εντολή του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, του ΦΡΑ. Βέβαια το θέμα αυτό εξακολουθεί να αποτελεί θέμα εθνικής κυριαρχίας, ε, αλλά παρόλα αυτά εγώ υπερψήφισα την έκθεση. Η κυρία Βυσνιεύσκα απουσιάζει, ο λόγος τον κύριο Χάραν έφυγε και αυτός, η κυρία Μάγερ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ήμασταν πολύ αργοί για να αντιδράσουμε σε αυτό την Ουγγαρία και το Συμβούλιο κατεπηγόντω θα πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία του άρθρου 7. Διότι έχουμε κοινέ ευρωπαϊκέ αξίε ελεύθερη δημοκρατία και έχουν σημασία. Θα πρέπει να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά του. Ένα πανεπιστήμιο υποχρεώθηκε να μείνει εκτό και δεν υπάρχει ακαδημαϊκή ελευθερία. Η ανεξαρτησία του δικαστικού κλάδου απειλείται και οι μειονότητε κακομεταχειρίζονται. Από πλευρά ηθική και στρατηγική δεν θα πρέπει να ανεχθούμε το λαϊκισμό τη άκρα δεξιά. Διότι αν δεν δράσουμε γινόμαστε συνένοχοι και μεταθέτουμε το κέντρο βάρους τη πολιτική. Το είδαμε στη γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε περί προσφύγων που κατακλείζουν την Ευρώπη, που έγινε ανεκτή και πήγε από τελικά αντί να είναι κάτι ακραίο έγινε μια κοινοτοπία και το βλέπουμε και στην ιστορία μας και βλέπουμε τι φρίκε που, στις οποίες καταλήξαν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο δεν, δεν λειτουργήσε ποτέ ο, ο καθησυχασμός εκείνων που προθούν αρχέ που μισούμε ε, έκθεση Χάλς για, για τη Λιθουανία και το ποινικό αντιδραστήριο. και Ο κ. Ζαμάσκη έχει το λόγο για τον αφοπλισμό του ποινικού αντιδραστήρα. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, καταψήφισα την έκθεση του συναδέλφου, όχι διότι δεν θα πρέπει να διαθέσουμε χρηματοδότηση για τον αφοπλισμό αυτής της πυρηνικής ε, εγκατάστασης, αλλά είμαι κατά το να επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, στι αρχέ τη και τι αποφάσει επί των πολιτών. Έχουν το δικαίωμα οι πολίτε να αποφασίζουν για τη μοίρα του. Και αυτό θα πρέπει να αντιπροσωπεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι στο πλευρό εκείνων που καταψήφισαν τη δικτατορία των Βρυξελών προ κάποιων ετών. Η Βουλγαρία έκανε το ίδιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με μη δημοκρατικό τρόπο επέβαλε την απόφασή της επί της Βουλγαρίας και της Λιθουανίας να απενεργοποιήσουν ε, πυρηνικούς σταθμούς ε, ηλεκτρικής ενέργειας. Ήταν σαφές από την αρχή ότι ε, αφοπισμός αυτών των εγκαταστάσεων ήταν κάτι ανόητο, κάτι αποτελεσμα... αναποτελεσματικό. Παρά τα αυτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε τη βούλησή της επί των δυστύχων κρατών μελών. Ευχαριστώ. Ο κ. Φαρία. Ευχαριστώ. Εγώ υπερψήφισα την έκθεση, γιατί θα πρέπει να παραπληστεί ο πυρηνοελεκτρικό σταθμό του Ιγναλίνα στη Λιθουανία. Γιατί εφαρμόζει παροχημένη τεχνολογία, παρακαταθήκη της Σοβιετικής Ένωσης και είναι με μεγάλη ευκαιρία να αποκτήσουμε ε, γνώσεις ε, για τον παραπλησμό τέτοιων πυρηνικών σταθμών και χρειάζονται επενδύσεις για το θέμα αυτό. Επίσης, ε, θα πρέπει να έχουμε εξαίρεση από την αρχαιορυπένη πληρώνει για τα ε, ραδιενεργά απόβλητα. Γιατί η Σοβιετική Ένωση πρώην επέβαλε στη Λιθουανία αυτό τον ε, πυρηνικό σταθμό και η πληρωμή των, της διάθεσης των ραδιενεργών αποβλήτων είναι άδικη και την υπερβολική για τη μικρή αυτή χώρα. Και γι' αυτό έχει πολύ ψηλό κόστος για την τεχνολογία του παροπλισμού. Θα πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε με βάση το, την Euratom την Λιθουανία και να προβλεφθούν σχετικές επενδύσεις για τον παροπλισμό του πυρηνικού σταθμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και ως πισω έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Υπερψήφισα την πρόταση Θεωρώ ότι είναι καλό ένα, μια επικίνδυνη πυρηνική μονάδα τη Σοβιετική εποχή να σταματήσει να λειτουργεί. Είναι προ όφελο και των Λιθουανών και των Ευρωπαίων. Σαν παιδί, θυμάμαι την έκρηξη του Τσερνόμπιλ που έγινε και που είχε μεγάλο αντίκτυπο και για τη χώρα μας. Η αμφισβήτηση αυτής της προτάσεω θα ήταν κάτι ανόητο. Πιστεύω ότι ήταν ορθή η απόφαση και είναι σωστό η Ευρωπαϊκή Ένωση να εμπλέκεται όσον αφορά την απενεργοποίηση αυτού του πυρηνικού σταθμού παρέχοντας ε, κατάλληλη χρηματοδότηση. Είναι καλό που διατηρούμε την αρχική αναλογία οικονομικής βοήθειας για τον αφοπλισμό αυτού του πυρηνικού σταθμού που είναι επικίνδυνος. Είναι θετική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή και για λόγους σαφώς ασφαλείας συμφώνησε να σταματήσει να λειτουργεί αυτός ο σταθμός όταν προσεχώρησε η Λιθουανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και χαίρομαι που ενεκρίθη αυτή η πρόταση. Ευχαριστώ. Προχωρούμε στην επόμενη έκθεση για την προστασία του προπολογισμού της Ένωσης σχετικά με το κράτος δικαίου στα, κράτος μέλη, κράτη μέλη. Κυρία Σόιντρομ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. βασικός στόχος του κανονισμού είναι κάτι με το οποίο συμφωνώ. Να πω όμως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει ένα μέσο στη διάθεσή της για να επιβάλλει κυρώσεις κατά κάποιας χώρας που λόγω συστημικών ελιμάτων ελλείψεων ε, στο δικαστικό τη σύστημα δημιουργεί προβλήματα και κινδύνους για, το οικονομικό, για τα οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Με κάποιες πτυχές διαφωνώ της διαδικασίας. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε στον τριμερή διάλογο να εντοπίσουμε τις λεπτομέρειες. Παρά κάποιες αντιρρήσεις, θεωρώ ότι αυτό είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ένα τέτοιο εργαλείο στη διάθεσή της. Ευχαριστώ. Η κυρία Μακοβέη έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κανονισμός προστατεύει τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τα κράτη-μέλη που δεν τηρούν το κράτος δικαίου δημιουργούν μεγαλύτερη ζημιά στα οικονομικά τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, εκεί που απειλείται η ανεξαρτησία του δικαστικού κλάδου και όπου οι αποφάσει λαμβάνονται αυθαίρετα ή παράνομα, συμπεριλαμβανομένων και των αποφάσεων των δημοσίων αρχών που δεν τιμωρούνται μαλλιανθασμένε και δεν διορθώνονται και εκεί όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες περιορίζονται, όπως και η ελευθερία των ΜΜΕ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πολλές αποφάσεις που λαμβάνονται δυστυχώς, όπως στη Ρουμανία, ε, είναι επιβλαβείς. Στις χώρες εκείνες που δεν τηρείται το κράτος δικαίου, κινδυνεύει το ευρωπαϊκό χρήμα. Και ο κανονισμός προβλέπει τη δυνατότητα παγώματος ή αναστολής της διαθέσεως πόρων και θα πρέπει η χώρα τότε να καταβάλει πληρωμέ από το δικό του προπολογισμό και δεν θα χρηματοδοτείται με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι ότου να καλύψει τα διάφορα κενά και προβλήματα. Ευχαριστώ, κύριο Τζαμπάφσκι, έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ καταψήφισα την έκθεση αυτή γιατί δεν πιστεύω ότι είναι σωστή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί το άρθρο 7 προβλέπει μια διαδικασία που συνιστά περαιτέρω γραφειοκρατικό άχθος. Και ουσιαστικά χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για να ε, καταπολεμηθούν οι πολιτικοί αντίπαλοι. Και δεν θα πρέπει να πληρώνει τα σπασμένα ευρωπαίες πολίτες γιατί σε τελική ανάλυση δικαιούχος των κονδύλων αυτών είναι οι πολίτες. Και είναι υποκρισία να χρησιμοποιούν το επιχείρημα τη παραβίαση του κράτου δικαίου, γιατί είναι σαφή τα παραδείγματα τη Πολωνία και τη Ουγγαρίας. Δεν θα πρέπει να υπερέχουν τα συμφέροντα της Δυτικής Ευρώπης έναντι των συμφερόντων των χωρών τη Ανατολική Ευρώπη. γιατί αυτό βλέπουμε και στο πακέτο κινητικότητας. Ότι τα συμφέροντα τη Δυτικής Ευρώπη υπερέχουν το, το συμφέρον της Ανατολικής. Αυτό οδηγεί σε ευρωσκεπτικισμό. Ο κύριο Ποσπίσιλ. Σας ευχαριστώ. Αφιταλαντεύτηκα για πολλή ώρα ε, να υπερψηφίσω ή να κρατήσω στάση αποχής. Τελικά ψήφισα αποχή. Απ' τη μια χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να προσπίσει τις αρχές και αξίες της και άρα και το κράτος δικαίου μεταξύ αυτών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά η συγκεκριμένη πρόταση δεν είναι κατά τη γνώμη μου πολύ καλή. Υπάρχουν πολλά επίμαχα ζητήματα εδώ. Όπω το επισήμανε και η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου. Και παρά τι προσπάθειες να αναβραθεί συμβαστική λύση, υπάρχει ακόμη το πρόβλημα τη νομική βάση που δεν έχει επιληθεί. Θα παρακολουθήσω και στη συνέχεια τη συζήτηση επί τη προτάσεω, αλλά θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι οθετούμε μια πρόταση που θα έχει ε, στέρεη νομική βάση, πάγια νομική βάση που θα πορεύει από το ενωσιακό δίκαιο. Και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί κάτι τέτοιο ως ε, επέκταση των ε, ιδρυτικών συνδικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυρία Ζαμπορσκά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συγκεκριμένη πρόταση έχει τρεις βασικές αδυναμίες. Πρώτον, η... δεν είναι δική Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόσφατα η Γαλλία ανακοίνωσε υπέρβαση των δημοσιονομικών ορίων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ εύκολα τη έδωσε εξαίρεση. Δεν υπάρχει η συμμεταχείριση της Γαλλίας και της Πολωνίας, για παράδειγμα, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, επειδή είναι πολύ γενικές και όριστε οι διατάξει ε, του κειμένου, δίνουν ε, λαβή για ε, διαφορετικές ερμηνείες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δίωξη των πολιτικών αντιπάλων. Επίσης, ε, με αντιστραμμένη ενισχυμένη πλειοψηφία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να προτείνει ε, ακυρώσεις που θα εφαρμόζονται αυτόματα εκτός και αν η ενισχυμένη πλειοψηφία αποφασίσει διαφορετικά. Ουσιαστικά δηλαδή το Συμβούλιο γίνεται δευτεροβάθμιο δικαστήριο ε, και με πολύ μικρές πιθανότητες επιτυχίας να ανατρέψει απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Περνάμε στο πρόγραμμα Φισκάλης για τη φορολογία. Κύριε Μακοβέη. Σας ευχαριστώ. Οι φορολογικές συμφωνίες που τυπικά δεν παραβιάζουν την νομοθεσία οδήγησε σε απώλεια φορολογικών εισόδων ε, πολλών δισεκατομμυρίων από το κοινοτικό και εθνικούς προϋπολογισμούς. Η φοροδιαφυγή, η φοροαποφυγή, οι διασυνοριακά εγκλήματα ή ξέπλυμα χρήματος επιτρέπουν ε, στις εθνικές αρχές, χάρη στο πρόγραμμα, να ανταλλάξουν πληροφορίες και τεχνογνωσία, ώστε να βρουν τους δράστες και να ανακτήσουν τα ε, φορολογικά έσοδα. Είναι σημαντικό να ανακτηθούν αυτά τα έσοδα και να ε, μην επιτρέψουμε τη συνέχιση τέτοιων εγκλημάτων. Η πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής θα πρέπει να παραμείνει προτεραιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδε μη, θα οδηγηθούμε στις κυρώσεις, όπως είχαμε και με την έκθεση Άρβαμα, λόγω της παραβίας του κράτους δικαίου. Και θα τιμωρηθούν οι πολιτικοί θύνοντες τελικά, γιατί δεν λαμβάνουν υπόψη το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών. Περνάμε στην έκθεση για το πρόγραμμα για τα δικαιώματα και τις αξίες. Η κυρία Σόιντροβα. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι, υπερψήφισα το πρόγραμμα για τα δικαιώματα και τις αξίες. Ε, το θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίζει τις δραστηριότητε των πολιτών. Θα πρέπει ο κόσμος να μπορεί να συναντάται, να γνωρίζει ο ένας τον άλλον, να υπάρχει επαφή μεταξύ κρατών μελών και να υπάρχει επαφή και σε περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο πόλεων όμως. Επίσης, υπερψήφισα και το θέμα των αξιών, το πρόγραμμα για την πρόθεση των αξιών που θα πρέπει να μεταφέρει χρήματα από τις περιφέρειες προς το κέντρο σε περίπτωση όπου ένα κράτος μέλος παραβιάζει το κράτος δικαίου. Δεν νομίζω ότι πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση όμως. Διότι είναι ένα οικονομικό πρόγραμμα το οποίο υποστηρίζει δραστηριότητες και δεν θα πρέπει να καθορίζει πολιτικά ζητήματα. Ευχαριστώ κύριο Ζαμπαύσκη, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν υποστήριξα την έκθεση αυτή του συναδέλφου για τα δικαιώματα και αξίες του συναδέλφου, του συναδέλφου Βαλέρο, διότι αυτό το μέσο τελικά παρεμβαίνει στα κυρίαρχα δικαιώματα των κρατών μελών. Επίσης είδαμε τι συνέβη στην Ουγγαρία και στην Πολωνία. Ε, παρεβιάζει την κυριαρχία των χωρών αυτών. Ε, προτείνω να έχουμε ένα νέο στόχο που θα σχετίζεται με το κράτος δικαίου και τις δημοκρατικές αρχές. Ε, διαφορετικά μέσα χρησιμοποιούνται όμως τώρα σε διαφορετικά επίπεδα μέσα τα οποία παραβιάζουν τα δικαιώματα κάποιων χωρών. Η Ρίστον Παρόδο, η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης που είναι ένα τέτοιο εργαλείο κανένα, καμία τέτοια υποκριτική προσέγγιση και μέσο δεν θα πρέπει να ενταχθεί στα προγράμματα αυτά για τις ε, αξίες και τα δικαιώματα. Ευχαριστώ κύριε Σπάλμερ. Ευχαριστώ κυρία Αντιπρόεδρε. Το πολιτικό χάος αυτής της εβδομάδας ε, ε, αφήνει δύο ομάδες ανθρώπων με αβεβαιότητα του πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω που ζουν και εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και πολίτε του Ηνωμένου Βασιλείου που ζουν σε κάτι με τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Γιατροί και νοσηλευτέ, κτίστε, υδραυλικοί, δάσκαλοι, ακαδημαϊκοί, δημόσιοι υπάλληλοι, επιχειρηματίε, ιδιοκτήτε επιχειρήσεων. Επίση πατεράδε, μητέρε, παππούδε, γιαγιάδε, αδελφέ, αδελφοί, φοιτητέ, μαθητέ. Αυτοί είναι πραγματικοί άνθρωποι. Δεν είναι μια αφηρημένη έννοια και αφηρημένα ζητήματα. Απευθύνω έκκληση λοιπόν προς το Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να επιλύσουν το θέμα αυτό για να διαφυλάξουν τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων ε, χωρίς καμία καθυστέρηση. Σας ευχαριστώ. Πάμε στην έκθεση Ο Κύριος Άνναν απουσιάζει. Η κυρία Άντερσον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπερψήφισα την έκθεση μαζί με την ευρύτερη πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η καθυστέρηση πληρωμέ υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχονται αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για τις μικρομεσαίε επιχειρήσεις, 85% των οποίων στον Ηνωμένο Βασίλειο δηλώνουν πως καταβάλλονται αργά οι αμοιβέ, ενώ 17% μιλούν για καθυστερημένε πληρωμές ακόμη και μετά τι 60 ημέρε που ορίζονται ω όριο για την προθεσμία υπερημερίας. Γι' αυτό λοιπόν ε, θεωρώ ότι έχει τεράστιο κίνδυνο, ενέχει ναι, τεράστιο κίνδυνο αυτό το πρόβλημα των ε, καθυστερημένων πληρωμών, τις οποίες αντιμετωπίζει η έκθεσή μου. Βέβαια, επιτρέπεται να συνεχιστεί με κάποιο τρόπο η καθυστέρηση. Γι' αυτό χαίρομαι που ζητούμε νομοθετική δράση και παρέμβαση όπου χρειάζεται για να υιοθετηθεί μια πιο αυστηρή στάση έναντι εκείνων που καθυστερούν να, πληρώσουν και ιδιαίτερα στις διαδικασίες των διαγωνισμών και άλλες αντίστοιχες οι οποίες σημαίνουν καθυστέρηση πληρωμών από δημόσιους φορείς για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενη έκθεση Τζιρόν για την διαφοροποιημένη ολοκλήρωση και το λόγο έχει ο κύριος Ελίμωβιτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ιδέα μια διαφοροποιημένη ολοκληρώσης δεν είναι καινούργια ιδέα. Την έχουμε στην ε, Τραπεζική Ένωση υπό όρους διαφορετικούς από ό,τι στο Σέγγεν, από ό,τι διαφορετικούς από ό,τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως τώρα φαίνεται κάποιοι μιλούν για μια διαφοροποιημένη ολοκλήρωση, εννοώντας ότι πρέπει κάποιες χώρες να ενωθούν περισσότερο, αφήνοντας, ε, βγαίνοντας έξω από αυτό το πνεύμα συνεργασίας. Έτσι λοιπόν και καθώς ε, ιδιαίτερα μεριμνό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να σταθώ κατά αυτής ε, της ιδέας, γιατί το να είναι κανείς μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης και το λέω αυτό παρότι είμαι επικριτικό, σημαίνει ότι πρέπει να είναι να, πάντα διατεθειμένος να κάνει συμβιβασμούς. Αυτό είναι μια δυναμία μας βεβαίως, αλλά και σημείο που μπορεί να κρυθεί και ως πλεονέκτημα. Και βεβαίως μαθαίνουμε ένας ε, από τον άλλον, μπορούμε να λύνουμε τα προβλήματα όλου του κόσμου μαζί. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ, αν δεν είμαστε όλοι μαζί, να αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριος Νέκοφ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η διαφοροποιημένη ολοκλήρωση είναι απλώς ένας ευμιστικός τρόπος για να ε, δικαιολογηθεί η σχάση του πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κατανομή των πολιτών σε κατηγορίες πρώτη, δεύτερη, τρίτη κτλ. Δηλαδή διπλά μέτρα και σταθμά εισάγονται. Είναι πολύ λυπηρό και επώδυνο για την πατρίδα μου αυτό που βλέπουμε. Ε, δεν είναι δυνατόν να προσπαθούμε να απαλείψουμε τα διπλά μέτρα και σταθμά στα τρόφιμα, αλλά να αφήνουμε την ε, ε, Βουλγαρία και τη Ρουμανία εκτός του Σέγγεν, γιατί όταν οι χώρες αυτές δεν αισθάνονται ισότιμες με τις άλλες, όπως οι πολίτες τους, παραδείγματι, δεν θα υιοθετήσουν, δεν θα ενστερνιστούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και οι άλλοι πολίτες. Πρέπει λοιπόν να μιλήσουμε για το θέμα αυτό έχοντας υπόψη πόσο χαμηλές είναι, χαμηλά και τα ποσοστά προσέλευσης στην κάλπη που είναι πάντα πολύ χαμηλό. Κύριο Σφαρία. Ευχαριστώ. Ψήφισε υπέρ γιατί θεωρώ ότι η διαφοροποιημένη ολοκλήρωση προβλέπει μια Ευρώπη που δεν λειτουργεί με την ίδια ταχύτητα. Και θα πρέπει να είναι συνταγματικό μέσο που θα εξασφαλίζει ελαστικότητα χωρίς να διακυβεύει το την ισότητα μεταξύ των πολιτών και το πολιτικό σύστημα. Θα πρέπει να, έχουμε, να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες των κρατών μελών να εφαρμόσουν αναπτυξιακέ πολιτικές χωρίς να δημιουργούμε Ευρώπες, Ευρώπη δύο ταχυτήτων και πολίτε πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Θα πρέπει επίσης να αποφύγουμε την αυτοεξαίρεση ή παραβίαση του πρωτογενούς δικαίου, γιατί κάτι τέτοιο διακυβεύει την κοινωνική συνοχή της Ένωσης. Δεν μπορούμε όμως να μιλούμε άσχημα για τι θεμελιώδεις αξίες και αρχέ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η λύθη δεν θα πρέπει να υπάγονται στη διαφοροποιημένη ολοκλήρωση. Στο μελλοντικό θεσμικό πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να ξεχνούμε τα πολιτικά, δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουμε τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά, οικονομικά και άλλα συμφέροντα. Δεν επιτρέπονται εξαιρέσει σε τέτοιου σημαντικά ζητήματα όπω είναι η καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Περάμε στην τελευταία έκθεση για τη στρατηγική έρευνα τη διαμεσολαβήτρια. Κυρία Εύη, το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το το κλειδί για να δώσουμε ένα νέο νόημα σε αυτή την Ευρώπη βρίσκεται στη νομοθεσία που υιοθετούμε σήμερα, που υιοθετήσαμε σήμερα και ονομάζεται διαφάνεια. Δεν μπορεί να συνεχίσει και κλεισμένον των θυρών να λαμβάνει αποφάσεις, να εκδίδει έγγραφα και να δίνει εντολές στους πολίτε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη από το 2018 ήταν σαφές ότι θα πρέπει να εξασφαλιστούν οι αρχές της διαφάνειας και τη αντικειμενικότητας σε κάθε, και της δημοσιότητα σε κάθε φάση των εργασιών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Ένα συγκεκριμένο μέτρο για να μπορέσει η Ευρώπη αυτή να γίνει κοινό σπίτι, κοινό οίκο όλων των Ευρωπαίων που θα υπερασπίστε τα δικαιώματά του, τις κοινωνικέ, τα κοινωνικά του δικαιώματα, θα αντιμετωπίζει τι αδικίες, θα ζει σε αρμονική σχέση με τον υπόλοιπο πλανήτη. Έτσι λοιπόν θέλουμε να έχουμε ένα παλάτι διαφανές, ένα παλάτι καθαρό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αγαπητοί συνάδελφοι, διακόπτουμε μέχρι τις 3.